being seen as the Mr. has taken on the mantle of Mr. Λοιπόν, ο, ε, ο κύριος Κράμερ μας υπενθυμίζει ότι έχει περάσει η ώρα. Ε, δηλώνω λοιπόν την έναρξη της συνεδρίασης. Θα, ήθελα να συγχαρώ τους Ισπανούς συνάδελφους, δεν βλέπω κανέναν. Οπότε τι να κάνω, να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου στους Ολλανδούς για το Μουντιάλ. Τέλο πάντων. Συμβαίνουν αυτά στον αθλητισμό, έτσι δεν είναι. Ε, πρώτο θέμα έγκριση ημερήσια διάταξη. Εγκρίνεται. Ναι. Σα ευχαριστώ. Στη συνέχεια έχουμε την έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης στις 21, 20, στις 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου. Εντάξει, έχετε κανένα πρόβλημα. Ευχαριστώ. Επόμενο θέμα. Κοινωνική διάσταση εσωτερική αγορά των αεροπορικών μεταφορών. Ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχουμε τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχετε το λόγο. Για 10 λεπτά περίπου. Και μετά θα σχολιάσουν τα μέλη της Επιτροπής μας. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα θυμάστε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμεύτηκε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την έγκριση ε, της αναθεώρησης ε, της αναδιατύπωσης της τρίτης δέσμης ε, Υπάρχει κάποιο τεχνικό πρόβλημα από ό,τι φαίνεται. Αν θα μπορούσατε να αρχίσετε ε, από την αρχή, λέει ο Πρόεδρο, σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα θυμάστε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε δεσμευθεί ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, κατά την αναδιατύπωση της, ε, του, της τρίτης δέσμης, αεροπορικής δέσμης του 1992 να παρουσιάσει ένα πανόραμα της κοινωνικής διάστασης της ιστορικής αγοράς στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών συγκεντρώνοντας την προσοχή της στις άμεσες επιπτώσεις ε, της εσωτερικής αγοράς επί των αεροπορικών μεταφορών ε, και βεβαίω ε, ε, χωρίς να ασχοληθούμε με τις ε, ε, οικονομικές συνέπειες. Το έγγραφο που έχετε μπροστά σας είναι καρπός μιας εργασίας που ενδεχομένως να κρίνεται ως μακροχρόνια. Φιλοδοξία μας όμως ήταν πρώτα απ' όλα να παρουσιάσουμε ποσοτικά στοιχεία όσον, στον τομέα της απασχόλησης, κυρίως για την εξέλιξη από το 1997 έως το 2007, αλλά ταυτόχρονα και κυρίως θα έλεγα να ε, υπάρξει μια ποιοτική ανάλυση των βασικών επιτευγμάτων και κοινωνικών διακυβευμάτων σε εσωτερική αγορά στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών. Λοιπόν, το έγγραφο αυτό όμω ε, έχει ε, περιορισμού και του συνειδητοποιούμε και εμεί ε, πρώτα απ' όλα. Να σα ομολογήσω λοιπόν ότι η απόκτηση των πληροφοριών που έχετε μπροστά σα δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερα εύκολο θα έλεγα. Υπήρξαν διάφορε πηγέ πληροφοριών Εργαστήκαμε ιδιαίτερα με τις διάφορες πηγές, είχαμε μερικά δεδομένα και έπρεπε να εμβαθύνουμε τις έρευνές μας για να ε, υπάρξουν ε, στατιστικά στοιχεία τα οποία να στέκουν κάπως. Σα πω λοιπόν αυτή εξ αρχή ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνειδητοποιεί την ανάγκη ε, επικαιροποίηση αυτού του εγγράφου και αυτών των στοιχείων και δεσμευόμαστε ε, ευθύ εξ αρχή προ την κατεύθυνση πληρωματικών μελετών. Όπω για παράδειγμα, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πρέπει να ληφθούν υπόψη οι συνέπειε τη οικονομική κρίση, τη πρόσφατη οικονομική κρίση, συνεχιζόμενη κρίση, στο συγκεκριμένο τομέα. Άρα λοιπόν δεν μπορούσε το συγκεκριμένο έγγραφο να λάβει υπόψη ε, τι συνέπειε τη κρίση. Τούτων λεχθέντων και παρόλους τους περιορισμούς αυτούς ε, θεωρούμε ότι είναι χρήσιμο και σας ευχαριστούμε κύριε Πρόεδρε που συμπεριλάβατε το έγγραφο αυτό στην ημερήσια διάταξη σήμερα. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε ευθύ εξ αρχή τον προβληματισμό και την ανταλλαγή απόψε με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ελπίζουμε να εμπλουτίσετε με τις απόψεις τη συζήτηση για αυτή την τόσο σημαντική πτυχή του τομέα των αεροπορικών μεταφορών. Τα αριθμητικά στοιχεία τα έχετε στο έγγραφο αυτό, τα είδατε άλλωστε. Να σταθούμε στο εξή, ότι καθόλου αυτό το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εξετάσαμε την απασχόληση στον τομέα των ε, ε, αεροπορικών μεταφορών, οι αεροπορικές εταιρείε ε, αυξάνονται κατά 6% το χρόνο και αυτό είναι πολύ σημαντικό. 25.000 εργαζόμενοι παραπάνω στον τομέα. Πράγμα που ε, θα μας επιτρέψει ενδεχομένως να καταλήξουμε σε ένα πρώτο συμπέρασμα, σε μια πρώτη ανάλυση τουλάχιστον, που έχει να κάνει με το γεγονός ότι η δημιουργία εσωτερικής αγοράς στο τομέα των αεροπορικών μεταφορών δεν οδήγησε σε ε, μείωση της απασχόλησης, τουλάχιστον συγκεκριμένο αυτό το τομέα, ενώ έγινε σε άλλους. προωθώντας την ανάπτυξη της εναέρειας κυκλοφορίας με νέες οδούς, με νέες εταιρείε, η κοινή αγορά ε, στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών όχι μόνο επέτρεψε τη σταθεροποίηση των θέσεων απασχόλησης, αλλά και τη δημιουργία δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Οι μελέτες ε, που διεξάγαμε έδειξαν ότι υπάρχει σαφώς ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στην ανάπτυξη της ε, ε, κυκλοφορίας, της κυκλοφορίας και στην εξέλιξη, της θετική εξέλιξη απασχόλησης. Επίσης μπορέσαμε να δούμε ότι η εσωτερική αγορά είχε αποτέλεσμα με την κατάσταση ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι εδώ δεν φαίνεται και το αποδεικνύουμε δεν ισχύει κάτι τέτοιο γιατί στην ουσία ε, ο βασικός παράγοντας για τη γεωγραφική κατανομή της απασχόλησης στο συγκεκριμένο τομέα είναι ο τόπος απογείωση και προσγείωση των αεροπλάνων. Έτσι. Ε, είναι προφανές αλλά δεν πρέπει να το ξεχνάμε και όπως και για κάθε άλλη ε, δραστηριότητα παροχής υπηρεσιών και εδώ υπάρχει ισχυρή συσχέτιση ανάμεσα στον τόπο παροχής υπηρεσίας και στον τόπο δημιουργίας ε, απασχόλησης. Με άλλα λόγια, οι εργαζόμενοι στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών βρίσκονται, και αυτό είναι φυσιολογικό, ε, στην ίδια ε, περιοχή με τον χρήστη, δηλαδή τον επιβάτη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και αν θα μπορούσα να προτείνω ένα τύπο, πρόεδρε, σε ζητώ συγγνώμη, οι αεροπορικές μεταφορές είναι ένα είδο ε, υπηρεσίας ε, ε αν θέλετε για να ε, αν μπορώ να το θέσω έτσι ε, να σας πω όμως κάτι άλλο και αυτό είναι πραγματικότητα η απασχόληση στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών στο σύνολό του εξελίχθηκε εξελίχθηκε διαφορετικά θα λέγαμε παρόλο που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι ένας, ένας ορισμένος ε, ε, ένας αριθμός επαγγελμάτων στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών δεν λαμβάνεται υπόψη γιατί γίνεται εξωτερική ανάθεση από τι ίδιες αεροπορικέ εταιρείε, όπω για παράδειγμα ε, η τροφοδοσία, το catering. Αλλά και εδώ και πέραν αυτής της συνολικής αντιμετώπισης του τομέα, σαφώς η εναέριος κυκλοφορία ε, και οι εναέρειες μεταφορές είναι αυτές που ε, σχετίζονται με την, ε, με την απασχόληση. Είτε πρόκειται για ολόκληρες τις αεροπορικές εταιρείε από την κορφή της πυραμίδας μέχρι τη βάση, είτε πρόκειται για εξωτερική ανάθεση μέρους των υπηρεσιών. Τώρα, όσον αφορά την ποιοτική εξέλιξη στον τομέα, τι συμπεράσματα μπορούμε να αντλήσουμε. Αυτό το οποίο μπορέσαμε να δούμε είναι ότι υπάρχουν ισχυρέ συνέπειες, σοβαρέ συνέπειε όσον αφορά ε, την διατήρηση και τη λειτουργία τη αγορά-εργασία στο συγκεκριμένο κλάδο. Πρώτα απ' όλα, επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια για κάτι το οποίο είναι σημαντικό και το οποίο έχει να κάνει με την ανάπτυξη παραγωγικότητας αλλά και με την ευελιξία ε, της εργασίας στο συγκεκριμένο τομέα. Συνολικά, ε, ο όγκος απασχόλησης ε, ε, ε, είχε θετική εξέλιξη με την εσωτερική αγορά, το είπαμε. Ταυτόχρονα όμως, και αυτό είναι αδιαφυσβήτητο, ο τομέας γνώρισε βαθιές αλλαγές ως προς τις συνθήκες εργασίας και αυτό συνδέεται και με την διαρθρωτική εξέλιξη που έχει να κάνει με το σύνολο της οικονομίας αλλά και με το θέμα του ανταγωνισμού στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών. Ανταγωνισμός που συνδέεται άμεσα φυσικά με την εσωτερική αγορά. Τώρα, όσον αφορά την εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων, που όπως είπα και πριν από λίγο, δραστηριότητες στο παρελθόν εντάσσονταν στην ενιαία, στην ενιαία δομή, όπως για παράδειγμα ε, η συντήρηση ε, ή η τροφοδοσία ε, σε σε διάφορες ενδιάμεσους σταθμούς, επίσης οι εταιρείες χαμηλού κόστους. Όλα αυτά οδήγησαν στην εξέλιξη στη βαθιά εξέλιξη της δομής της απασχόλησης. Και κατά το χρονικό διάστημα 1997 έως 2007 πράγματι παρατηρήσαμε διαδικασίες πολύ σημαντικές αναδιάρθρωσης και εξωτερικής ανάθεσης ε, τμήματος υπηρεσιών και όλα αυτά είχαν επιπτώσει στο σύνολο των ε, επαγγελμάτων που εμπλέκονται σε αεροπορικές μεταφορές. Άρα λοιπόν ε, η παραγωγικότητα, και πρέπει να πούμε ότι η παραγωγικότητα αυξήθηκε σε σημαντικό βαθμό. Αυτό πρέπει να το σημειώσουμε και δεν το ξεχνάμε. Ένα παράδειγμα να σας δώσω. Ο μέσος αριθμός ε, απασχολούμενος στον τομέα που, που χρειάζεται ε, μια αεροπορική εταιρεία για να μεταφέρει χίλιους επιβάτες μειώθηκε κατά 36% τα τελευταία 10 χρόνια. Βλέπετε λοιπόν σημαντική ανάπτυξη της παραγωγικότητας. Δεύτερη πτυχή. Ε, η ανταγωνιστική πίεση που μεταφράζεται σαφώς σε, σε προσπάθεια για επίτευξη ε, μεγαλύτερη ευελιξία. Αυτό ισχύει σε όλου του κλάδου και στο τομέα των αεροπορικών μεταφορών. Ε, ισχύει ο ίδιο κανόνα. Για παράδειγμα, η αύξηση του αριθμού των συμβάσεων μερική απασχόληση στο τομέα αεροπορικών μεταφορών είναι σημαντική και αφορά πλέον το 20% των απασχολούμενων ήταν 20% το 2006. Διπλάσιος ο ρυθμός έναντι των απασχολούμενων το 1997. Άλλο θέμα, ε, διάρθρωση του μισθού και των αποδοχών. Και εδώ έχουμε εξελίξεις. Ε, και όλο και σε μεγαλύτερο βαθμό μεταβλητές αποδοχές. Ε, πρώτη ποιοτική εξέλιξη και η δεύτερη έχει να κάνει με τα διακυβεύματα της εξέλιξης της απασχόλησης σε διεθνικό επίπεδο. Δεν πρόκειται για ιδιαιτερότητα του τομέα των αεροπορικών μεταφορών, αλλά σαφώς αυτή η διεθνική πτυχή στις συγκεκριμένες δραστηριότητε είναι κάτι το πολύ σημαντικό. και, στην αεροπορία, και στις αεροπορικές μεταφορές όπως και στους άλλους οικονομικούς ε, κλάδους ε, ε, το, το, εδώ πρέπει να μιλήσουμε για ένα κοινό, για κοινά πλαίσια που έχουν να κάνουν με την κοινωνική προστασία. Υπάρχουν βεβαίως ιδιαίτερα πρότυπα τα οποία ισχύουν στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών και τα οποία ε, προσδιορίζονται κυρίω για λόγου ασφαλείας. Και αυτά έχουν σημαντικές συνέπειες στι συνθήκε εργασία των απασχολούμενων στον αλόγο τομέα. Όμως, θα πρέπει να σημειώσουμε ταυτόχρονα ότι υπάρχουν εδώ στοιχεία ε, βασικά που αφορούν τις συνθήκες απασχόλησης και εργασίας ε, και τα οποία ε, εξακολουθούν να στηρίζονται σε εθνική βάση. Η ανάπτυξη λοιπόν του διεθνικού χαρακτήρα ως προς τις αυτές πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι αποτελεί μια, εξακολουθεί να αποτελεί μια πρόκληση για το συγκεκριμένο κλάδο. Και άλλωστε αυτό το ζήτημα το οποίο ε, απασχολούσε, ε, υπήρχε στο επίκεντρο των ανησιών του Κοινοβουλίου, ο, ε, συζητήθηκε όταν έγιναν οι διαπραγματεύσεις της αναθεώρησης του, του, του, της τρίτης ε, δέσμης αεροπορικών μέτρων που οδήγησε στην έγκριση τον Νοέμβριο 2008 του κανονισμού 1008. Πρόκειται λοιπόν για μια προβληματική, αναφέρομαι λοιπόν στην διεθνική απασχόληση που ε, ε, αποκτά όλο και πιο περίπλοκο χαρακτήρα λόγω των πρόσφατων εξελίξεων. Η δημιουργία τη ιστορικής αγορά στον τομέα των ευρωπαϊκών μεταφορών επίση έχει και μια άλλη συνέπεια ω προ την εξέλιξη της ευρωπαϊκή διάσταση των εταιριών και ε, τη ε, του τομέα ας σκεφτούμε τις συμφωνίες ε, που ισχύουν πλέον μεταξύ της Air France και της KLM που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ίδιο και αύριο με την ε, Iberia και την British Airways όλα αυτά έχουν ε, επιπτώσεις και όσον αφορά την ανάπτυξη εταιριών χαμηλού κόστους. Όλα αυτά βεβαίως έχουν άμεση σύνδεση με την απασχόληση του στον τομέα και με την εξέλιξη της απασχόλησης. Η εξέλιξη αυτών των διεθνικών επιχειρήσεων που ε, έχουν την έδρα τους σε πολλά κράτη-μέλη με προσωπικό το οποίο ε, προσλαμβάνεται ή εργάζεται σε διάφορες χώρες. Αυτές λοιπόν οι ιδιαίτερες συνθήκες δημιουργούν στο συγκεκριμένο τομέα ε, μια προβληματική που βρίσκουμε άλλωστε και σε άλλους τομείς παροχής διεθνικών και πολυεθνικών υπηρεσιών. Αυτό που πρέπει να σημειώσουμε είναι ότι οι συνθήκε απασχόληση και εργασία που αφορούν στου εργαζόμενου του ε, τομέα των αεροπορικών μεταφορών εξακολουθούν λοιπόν να προσδιορίζονται κατά βάση ε, από τα εθνικά πλαίσια. Και αυτό ισχύει κυρίω ε, ω προ τα κοινωνικά πρότυπα. Τα πολύ σημαντικά, όπως για παράδειγμα αυτά που αφορούν τις άδειες, τις εισφορές στο Ταμείο Συνταξιοδότησης, ε, τους ελάχιστους μισθούς όταν προβλέπεται ελάχιστη αμοιβή, στην εκπροσώπηση των εργαζομένων ή στα δικαιώματά τους σε περίπτωση απόλυσης. Να προσθέσω ότι η βέλτιστη και ισότιμη ε, λειτουργία της εσωτερικής αγοράς απαιτεί ένα ελάχιστο επίπεδο ε, κοινωνικών κανόνων που να ισχύουν και για τον τομέα των αεροπορικών μεταφορών, κυρίως όσον αφορά το υπτάμενο προσωπικό. Και αυτό προσπαθούμε να πετύχουμε άλλωστε. Θα, να σας υπενθυμίσω την οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων, η οποία ε, επιφέρει ε, ορισμένε εγγύησει προ του ε, εργαζόμενου που αποτελούν αντικείμενο προσωρινή απόσπαση σε ένα άλλο κράτο μέλο, σε ένα κράτο μέλο δηλαδή διαφορετικό από αυτό στο οποίο συνηθίζουν να εργάζονται, έτσι ώστε αυτοί οι απασπόμενοι εργαζόμενοι να ωφελούνται από ένα ελάχιστο σκληρό πυρήνα δικαιωμάτων που θα πρέπει να σέβεται η χώρα υποδοχής. Και έχουμε μάλιστα και πρόσφατη νομολογία από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η Viking Line, η Laval για παράδειγμα, αυτές οι υποθέσεις όπου φαίνεται ότι υπάρχουν δυσκολίες όσον αφορά την ε, ε, υιοθέτηση και την υλοποίηση αυτής της οδηγίας και πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τη συμφιλίωση δύο κατηγοριών θεμελιωδών δικαιωμάτων, των κοινωνικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων που απορρέουν από την εσωτερική αγορά και του δικαίου που απορρέει από την εσωτερική αγορά. Προσπαθούμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτή τη δυσκολία και έχουμε δεσμευτεί προ την κατεύθυνση αυτή, λαμβάνοντα και μία σειρά από πρωτοβουλίε για τη βελτίωση τη ε, υλοποίηση αυτή τη τόσο σημαντική οδηγία που αφορά στην απόσπαση των εργαζομένων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει μια πρωτοβουλία, νομοθετική πρωτοβουλία ε, την οποία θα, θα υποβάλει του χρόνου έτσι ώστε να διευκρινιστούν στο μέτρο του δυνατού βεβαίω οι συνθήκε υλοποίηση και εφαρμογή τη συγκεκριμένη οδηγία που αφορά την ε, απόσπαση των εργαζομένων. Ένα άλλο πιο πρόσφατο παράδειγμα αφορά ε, τον κανονισμό 593 ε, που αφορά ε, τις συμβασιακές υποχρεώσεις ε, είναι ο κανονισμός ε, Ρώμη 1 ε, που προβλέπει ότι οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να στερούνται των επιτακτικής φύσεων διατάξεων του κράτους μέλους το οποίο, το τονίζω, ή από το οποίο, ε, ε, ε, στο οποίο δηλαδή ασκούν συνήθως επαγγελματικές δραστηριότητες. Άρα δηλαδή και εδώ πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη εφόσον ο συγκεκριμένος κανονισμός έχει συμπεριλάβει τις ιδιαίτερες συνθήκες της, της κινητής εργασίας θα λέγαμε και προκειμένου το άρθρο 8. Αλλά αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο τα ευρωπαϊκά όργανα αλλά και τα εθνικά όργανα θα πρέπει ε, να σταθούν ιδιαίτερα και να επαγρυπνούν ιδιαίτερα θα έλεγα. Και τέλος, ε, τελευταία παρατήρηση, αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, από όλα αυτά τι πρέπει να κρατήσουμε αν θέλετε ε, και, πώς, και τι πρέπει να δούμε από το πρίσμα του κοινωνικού διαλόγου πρόκειται βεβαίω για μια ιδιαιτερότητα τη εσωτερική αγορά, ενιαία αγορά και κυρίω ενιαία αγορά στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών. Το γεγονό δηλαδή ότι επιτρέπεται στι αεροπορικέ εταιρείε να γίνουν ευρωπαϊκέ εταιρείε, ενώ ο κοινωνικό διάλογο ίσω ε, ε, δεν προβλέπει τι ίδιε διευκολύνσει, βεβαίω. Τούτου λεχθέντο, πολλοί μεταφορεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο και οι εργαζόμενοι τους έχουν αξιοποιήσει τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα ε, που ε, προβλέπει η 9445 ε, έτσι ώστε να δημιουργηθούν αυτά τα επιχειρησιακά συμβούλια τα οποία, στα οποία συγκεντρώνονται οι εκπρόσωποι όλων των εργαζομένων της επιχείρησης τώρα με, ε, με διεθνική μορφή αν θέλετε ε, στα διάφορα κράτη-μέλη. Και μέσω των οργάνων αυτών οι ε, εργαζόμενοι ενημερώνονται και, και, διαβουλεύονται με την, με την εργοδοσία όσον αφορά τις σημαντικές αποφάσεις που λαμβάνονται σε επίπεδο επιχείρησης και που ενδεχομένως μπορεί να επηρεάζει τους εργαζόμενους αυτούς. Θα έλεγα ότι η ανάγκη διεθνικής διαπραγμάτευσης κυρίως σε, θέματα, σε περίπτωση αναδιάρθρωσης η ανάγκη αυτή προκύπτει και με, ε, με τον όλο και αυξανόμενο αριθμό εταιριών και επιχειρήσεων που καταλήγουν σε συμφωνία παρά την απουσία νομικού πλαισίου σε συγκεκριμένο τομέα. Λοιπόν, εμείς σας λέω ότι υποστηρίζουμε αυτές τις εξελίξεις και αυτές τις συμφωνίες με διάφορες πρωτοβουλίες ε, και έχουμε δημιουργήσει και μια ομάδα εργασίας για να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο ε, γίνονται όλα αυτά, χωρίς να αποκλείεται μία ημέρα ενδεχομένως να υπάρξει ένα προαιρετικό νομικό πλαίσιο το οποίο θα συμπεριλαμβάνει κατά κάποιο τρόπο και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να αναπτύσσονται οι συμφωνίες αυτές και ε, πώς θα εμπλέκονται και οι εργαζόμενοι συμφωνίες αυτές. Γενικότερα, και εδώ θα τελειώσω κύριε Πρόεδρε, μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι η ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα γιατί οι συμφωνίες ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους θα μπορούσαν να αναπτυχθούν και, σε, ε, και στην κλίμακα ολόκληρου του τομέα των εμπορικών μεταφορών. Μην ξεχνάτε ότι η βασική δυσκολία του διαλόγου αυτού εξαρτάται από την αντιπροσωπευτικότητα των μερών και από την διαπραγματευτική εντολή που διαθέτουν. Ένα και μόνο παράδειγμα να σας δώσω για το θέμα αυτό, το οποίο όμως είναι σημαντικό. Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία που αφορά ε, την διαχείριση του χρόνου εργασίας του κινητού του αποσπόμενου προσωπικού στι αεροπορικέ μεταφο... στις αεροπορικές μεταφορές που, που ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 2000, 2000. Ε, το άρθρο 155 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσφέρει ε, τα επαρκή πλαίσια για ε, τέτοιου είδους διαπραγματεύσεις. Κύριε Πρόεδρε, αυτά ήθελα να σας πω. Τελειώνω εδώ. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Θέλησα πέραν μιας στήρας ε, και μηχανικής ε, ε, παρουσίας των δεδομένων που έχετε μπροστά σας και που το λέω για άλλη μια φορά ότι είναι μερικής φύσεως ατελή και θα πρέπει να επικυρωποιηθούν. Προσπαθήσαμε λοιπόν να χαράξουμε μια προοπτική όσον αφορά τα στοιχεία που είναι ποιοτική φύσεως και τα οποία είναι σημαντικά όταν θέλουμε να μιλήσουμε για την ενιαία αγορά στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών και για την εξέλιξή της από το 1997. Σας ευχαριστώ λοιπόν όλους για την προσοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Γκρός για το ΕΛΚ. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την παρουσίαση που έγινε. Για μένα ήταν αρκετά σαφής. Πιστεύω ότι είναι και σημαντική, καθώς Νομίζω ότι το θέμα αυτό αφορά όλους τους τομείς των μεταφορών. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τίθεται σε όλους τους τομείς των μεταφορών. Έτσι λοιπόν καλό θα ήταν να μπορούμε να έχουμε και παρόμοια ανάλυση και στις άλλες μεταφορές, θαλάσσιες, χερσές κτλ. Τώρα, ενή αγορά. Φυσικά η ενιαία αγορά έχει τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της. Αυτά που θα ήθελα να προσδιορίσω τώρα από την πλευρά του ΕΛΚ ήταν ότι τέτοιες αναλύσεις δεν θα πρέπει να οδηγούν σε λανθασμένα συμπεράσματα. Δηλαδή ότι η απελευθέρωση θα πρέπει να οπισθοχωρήσει γιατί έχουμε αρνητικές επιπτώσεις. Νομίζω ότι απλώς θα πρέπει να τα διορθώσουμε αυτά τα πράγματα όπως έγιναν σε κάποιες προτάσεις. Έτσι μπορούμε να πάμε παραπέρα, να αυξηθεί η απασχόληση, πολύ καλό. Αυτό αναμένουμε και από την ανοιχτή αγορά, αλλά επίση αναμένουμε όχι απλώ να υπάρχει αύξηση των θέσεων απασχόληση, αλλά να έχουμε και ποιοτικέ θέσει απασχόληση. Ε, θα πρέπει να πληρούνται κάποια κριτήρια για αυτέ τι ποιοτικέ θέσει απασχόληση. Νομίζω ότι έχουμε λάβει για κάποια κριτήρια τα κατάλληλα μέσα, ενώ για κάποια άλλα κριτήρια δεν τα έχουμε. Τώρα, για ε, τα κριτήρια που έχουμε τα μέσα, νομίζω ότι η μεταφορά στην ιστορική νομοθεσία των κρατών μελών ε, υπάρχει, έχουμε υφιστάμενη νομοθεσία και για μένα αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί νομίζω ότι θα είναι καταστροφικό να ανοίξουμε μια αγορά και να έχουμε ρύθμιση σε κάποιο τομέα και μην υπάρχει σωστή εφαρμογή από ορισμένε χώρε. Τώρα το δεύτερο είναι ότι στα μέσα που έχουμε υπάρχουν σε άλλα η κατάρτιση και νομίζω ότι η κατάρτιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ε, σε πλαίσιο ε, διεθνού, διεθνές ε, θα πρέπει να υλοποιείται αν μέσω πρόθεσμα ε, προκαλεί, ε, μάλλον δημιουργεί επισφαλής θέσεις εργασίας, ε, τότε δεν θα έχουμε ούτε ποιοτικέ θέσεις απασχόλησης ούτε θα πληρούνται οι προϋποθέσεις τη ασφάλεια. Αυτό είναι ένα πρώτο ερώτημα λοιπόν που θέλω να θέσω στην Κομισιόν σε ό,τι αφορά την αναθεώρηση των γενικών γραμμών. Θα το προσεγγίσουμε αυτό το θέμα, γιατί εμείς προσπαθήσαμε να έχουμε καλύτερη αγορά, αλλά δημιουργήσαμε πιο επισφαλείς συμβάσει σε ορισμένα αεροδρόμια και από την άλλη λέμε ότι ναι, ισχύει η εθνική νομοθεσία, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε ότι σε ορισμένα αεροδρόμια έχουμε ε, πάρα πολλές ε, διαφορετικές ε, συνθήκες απασχόλησης. Αυτό, αυτή είναι η δεύτερη δέσμη ερωτήσεων. Τρίτη τώρα πέρα από τις εταιρείε χαμηλού κόστους, low cost, ε, γιατί όπως είναι λογικό μάλλον θα προέρθει και χαμηλός μισθός από αυτές, έχουμε και τις παραδοσιακές εταιρείε, οι οποίες αναπτύσσονται προ δύο μεγάλα μονοπόλια κατά την άποψή μου. Έτσι λοιπόν στην Ευρώπη αυτή προσπαθούμε να βγούμε από τα μονοπόλια τα κρατικά, όμως δεν έχω την εντύπωση ότι στις αερομεταφορές ε, θέλουμε να προσεγγίσουμε ιδιωτικά μονοπόλια. Ίσως θα ήταν ενδιαφέρον η Κομισιόν να μας εξηγήσει το βάσιμο αυτών των ε, συνασπισμών που δημιουργούνται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε διεθνές επίπεδο και να δούμε αν επιτρέπεται η ύπαρξη πραγματικού ανταγωνισμού ή αν υπάρχει κίνδυνος να έχουμε ένα μεγάλο μονοπόλιο, το χάρη εφενός και να έχουμε τις εταιρείε υψηλού και αφετέρου τις εταιρείε χαμηλού κόστους. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα. Τώρα το τελευταίο θέμα αφορά αυτή την απόσπαση των εργαζομένων. Πολλές φορές εγώ ε, με το θέμα και έχουμε τη σχετική νομοθεσία. Πώς μπορεί να εφαρμοστεί εδώ σωστά η σχετική νομοθεσία. Το θέτω αυτό και στο πλαίσιο των διεθνών αερομεταφορών. Ως βουλευτές νομίζω ότι πολύ συχνά τίθεται ερωτήσεις, πρέπει να αντιμετωπίσουμε ερωτήσεις του τύπου εργάζομαι ε, στην τάδε χώρα, ενώ ζω, ζούσα σε μια άλλη χώρα και πρέπει να δούμε ποια νομοθεσία ισχύει, αν θα πρέπει να ισχύσει η οδηγία για την απόσπαση και αν ναι, πώς και πώς υπάρχει δυνατότητα ελέγχου, αν υπάρχουν μέσα ελέγχου. Γιατί απλώς το να πούμε ότι έχουμε μια οδηγία για την απόσπαση των εργαζομένων που εφαρμόζεται για τους εργαζομένους, αλλά να ξέρουμε ξέρουμε αφετέρου ότι δεν ελέγχεται και ούτε είναι δυνατόν να εφαρμοστεί, τότε δεν θα έχουμε κανένα θετικό αποτέλεσμα. Απλώς εφησυχαζόμαστε. Αυτές τις δέσμες ε, ερωτήσεων είχα για την ανακοίνωση αυτή. Σας ευχαριστώ για την παρουσίαση. Ευχαριστώ πολύ. Κύριος Ντράι. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω την Κομισιόν για την εισαγωγή αυτή και για την έκθεση. Νομίζω ότι το έγγραφο παρουσιάζει πολύ καλά την κατάσταση, αλλά θέτει και μια σειρά ερωτήσεων. Από ό,τι φαίνεται δεν έχουμε όλα τα δεδομένα. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διασφαλίσει στο μέλλον ότι όταν ε, μιλάμε για στατιστικά στοιχεία θα έχουμε σωστά και πλήρη δεδομένα. Δεν αναφέρομαι μόνο σε αυτό το φάκελο, αλλά και σε άλλους φακελούς που έχουν να κάνουν με τις μεταφορές ή στατιστικές. Φαίνεται να είναι συνεχές ε, πρόβλημα που μας δυσκολεύει να εξαγάγουμε συμπεράσματα. Είδαμε την ε, δεδομένη αύξηση στο τομέα. Είχαμε 40% αύξηση στον αριθμό των επιβατών στις κάτω χώρες. Όμως υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών. Σε ορισμένε χώρες είδαμε μείωση, ενώ σε άλλες είδαμε πολύ ταχεία αύξηση. Και όπως είπε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν στην εισαγωγή του, Επίσης είδαμε μεγάλη αύξηση στην ευελιξία και διπλασιάστηκε και ο αριθμός των βραχυπρόθεσμων συμβάσεων. Επίσης, ε, είδαμε να υπάρχουν και διαφορές μεταξύ των υποτομή. Ε, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των επισκευών, παραδείγματο χάρη, είδαμε ότι το επίπεδο της απασχόλησης παρέμεινε σταθερό παρά το ότι έχουμε 40% περισσότερους ταξιδιώτε. Ε, και αυτό σημαίνει ότι υπήρξε πολύ μεγάλη πίεση για μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Όμως, εγώ νομίζω ε, ότι αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει και μεγαλύτερη βιλξία από την πλευρά των εργαζομένων και στον τομέα αυτό των αποσκευών φαίνεται να έχουμε φτάσει στα όρια. Και ίσως έχει έρθει η κατάλληλη στιγμή να δούμε την ανάγκη προστασίας των εργαζομένων. Σε ό,τι αφορά τώρα τη συντήρηση των αεροσκαφών, δεν έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες για τον τομέα αυτό. Αναρωτιέμαι αν ε, έχει γίνει ε, εξωτερική ανάθεση για τη συντήρηση των αεροσκαφών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η εντύπωσή μου αλλά δεν υπάρχουν σχετικά στοιχεία στο έγγραφο. Τώρα για τον ενέργειο έλεγχο, τον έλεγχο της αερίου κυκλοφορία. Εδώ πρέπει να έχουμε προσωπικό με υψηλή εξειδίκευση, αλλά δεν έχουμε σαφή ιδέα σε σχέση με τον αντίκτυπο των σημερινών μεταρρυθμίσεων του ΣΕΖΑΡ, των νέων τεχνολογίων του ενιαίου Ευρωπαϊκού Ουρανού. Μπορείτε να μα δώσετε κάποιε ενδείξει για το τι πιστεύετε, για το ποιο μπορεί να είναι ο αντίκτυπο αυτών των αλλαγών σε αυτό το τομέα. Επίσης, Έχουμε και το σημαντικό ερώτημα ποια κοινωνικά πρότυπα πρέπει να ισχύουν για τις ε, διεθνείς αεροπορικές εταιρείες. Εδώ υπάρχει κίνδυνος τρέβλωσης του ανταγωνισμού. Αν οι αεροπορικέ εταιρείε ε, προσπαθούν να προσλάβουν προσωπικό σε χώρε όπου αυτό κοστίζει φθηνότερα, φυσικά αυτό δεν ισχύει για όλε τι κατηγορίε του προσωπικού, αλλά υπάρχει κίνδυνο τρέβλωση του ανταγωνισμού εδώ και φυσικά και κοινωνικού ντάμπινγκ. Έτσι λοιπόν νομίζω ότι θέσατε την ερώτηση αλλά δεν μας δώσετε απάντηση. Υπογραμμίσατε τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου ε, στα πλαίσια των εταιρεών. Νομίζω ότι όλοι είμαστε υπέρ αυτού. Ταυτόχρονα όμως δεν φαίνεται να προτείνεται ότι οι εργοδότες θα πρέπει να υποχρεούνται να, να ε, παρέχουν ένα οργανωτικό πλαίσιο. Δεν υπάρχει τέτοιο πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο θέμα αυτό θα ήθελα να σας ενθαρρύνω να προσπαθήσετε να βελτιώσετε την κατάσταση. Ίσως ε, στο μέλλον να διαρευνήσουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε κάποιο νομοθετικό πλαίσιο έτσι ώστε να ε, στηρίξουμε και να πλαισιώσουμε τις διάφορες πλευρές του κοινωνικού διαλόγου αυτό θα πρέπει να είναι μία μέγιστη προτεραιότητα κατά την άποψή μου. Ένα άλλο θέμα που δεν έχει απαντηθεί σαφή, σαφώς, θέλω να ρωτήσω. Τι πρωτοβουλία σκοπεύει να, να πάρει η Κομισιόν. πέραν των ε, τομέων ε, όπου έχει αφαιτηθεί η νομοθεσία. Δηλαδή, ποιες νέες πρωτοβουλίες αναμένεται να αναλάβει η Κομισιόν ε, σε ό,τι αφορά τους κανόνες ε, για την ε, κοινωνική προστασία στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ για τους λιμπήρους, κυρία Μάσνερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστούμε και εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίαση που μας έκανε εδώ. Πράγματι, θα πρέπει να δοθούν κάποιες απεραιτέρω διευκρινήσεις ε, φυσικά, ε, καταρχήν ε, χαιρετίζουμε την ενιαία εσωτερική αγορά. Αποτελεί ένα κεκτημένο για την Ευρώπη. Είναι κάτι το οποίο είναι προ όφελο όλων μα και θέλουμε να το διατηρήσουμε. Θα πρέπει όμω να εξετάσουμε πώ λειτουργεί η εσωτερική αγορά, πώ έχει διαρθρωθεί και αν είναι πραγματικά κοινωνική αγορά. Εγώ προέρχομαι από τη Γερμανία και στη Γερμανία λέμε συνέχεια ότι θα πρέπει να βασιζόμαστε στι αρχέ τη κοινωνική οικονομία τη αγορά. Ναι, λοιπόν, ναι στην ανταγωνιστική αγορά, αλλά να υπάρχουν και σωστέ κοινωνικέ προσφορέ, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τι θέσει εργασία και ούτω καθεξής. Έχω και κάποια πιο συγκεκριμένα ερωτήματα. Σε ό,τι αφορά του ελέγχου, θα αναφερθεί και ήδη από, ρωτήθηκε ήδη από τον κύριο Ραντό, δηλαδή το πώ έχουν τα πράγματα ε, για του ε, αρμόδιου ε, για τη συντήρηση των αεροσκαφών και από εκεί και μετά. Ένα ακόμα ζήτημα το οποίο έχει συζητηθεί επανειλημμένα είναι ε, η μισθή και γενικά η κοινωνική ασφάλιση ε, του προσωπικού το οποίο είναι αρμόδιο για τους ελέγχους ασφαλείας ε, στις πύλες των αεροδρομίων. Ε, πολύ συχνά αναφέρεται ότι υπάρχουν κάποιες ελλείψεις σε ό,τι αφορά ακριβώς αυτό το προσωπικό ε, γιατί δεν υπάρχει σωστή ε, αμοιβή για αυτά τα πρόσωπα. Αλλά από την άλλη πλευρά οι επιχειρήσεις που είναι αρμόδιες για τη διαχείριση των αεροδρομίων λένε ότι δεν μπορούν να δώσουν υψηλότερους μισθούς, γιατί κάτι τέτοιο θα είχε επιπτώσει στι ίδιε τι τιμέ των εισιτηρίων. Άρα λοιπόν σας ρωτώ τι ακριβώς θα κάνουμε σε σχέση με αυτό το προσωπικό. μετά μα είπατε η ε, πως ο αριθμός ή το, ε, το ποσοστό των, ε, της απασχόλησης των θέσεων εργασία μερικής απασχόλησης αυξήθηκε από το 10% στο 20% κυρίω έχουμε να κάνουμε με γυναίκε εδώ παρά με άντρε και έχουμε να κάνουμε κυρίω με πρόσωπα τα οποία θα ήθελαν να έχουν πράγματι πλήρη απασχόληση. Είναι περισσότερο κοινωνικού χαρακτήρα αυτέ τα ζητήματα, προφανώ, αλλά επειδή αναφερθήκατε και εσεί στην κοινωνική διάσταση, ε, τα θίγω. Ε, ειδικά και εν ώψη τη ε, τροποποίηση ε, τη ε, συνθήκη. Έχουμε δηλαδή αναφορά σε ό,τι αφορά κάποια συμβόλαια εργασία που είναι για πολύ μικροχρονικό διάστημα και προφανώ δεν είναι κάτι το οποίο επιθυμούν υποχρεωτικά οι εργαζόμενοι. Συχνά, βέβαια, κάτι τέτοιο αποτελεί τη μοναδική δυνατότητα για τη δημιουργία θέσεων εργασία από την πλευρά των εργοδοτών. Τώρα, αναφερθήκατε στο ζήτημα των εθνικών αρμοδιοτήτων σε ό,τι αφορά την ε, κοινωνική ασφάλιση. Από τη μία πλευρά, ε, στο πλαίσιο τη ε, ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη, θέλουμε να λάβουμε υπόψη μα τέτοια ζητήματα, για παράδειγμα, και να δούμε πώ κάποιο από την Ισπανία, ο οποίο εργάζεται στην Ιταλία, μπορεί να έχει μια σωστή ασφάλιση και το πιο δίκαιο θα ισχύει, αλλά το ερώτημα που θέτουμε εμείς είναι εσείς από τη δική σας πλευρά θεωρείτε πως θα πρέπει να επιτευχθεί περιττέρω προσέγγιση μεταξύ των εθνικών ε, νομοθεσιών. Εμείς δηλαδή ε, έχουμε ε, περισσότερο βασιστεί εδώ στη μέθοδο του ελεύθερου συντονισμού και όχι σε πραγματική εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών. Θέλετε λοιπόν να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Από εκεί και μετά, ε, στην κοινωνική διάσταση ε, της απασχόλησης ε, καταλέγονται και οι προσφορές περαιτέρω επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης. Πώς έχουν τα πράγματα στη σχέση λοιπόν με την επαγγελματική κατάρτιση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κράμερ του έχει το για τους πράσινους. Ευχαριστούμε και εμείς για αυτή την παρουσίαση. Το ζήτημα της κοινωνικής Ευρώπης ε, θέτει το ζήτημα της ε, λανθασμένης αν θέλετε οικοδόμησης ε, της Ευρώπης. Δηλαδή βασίστηκε αμυγός σε οικονομικά κριτήρια δημιουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά προσπαθούμε όλο ένα και περισσότερο να συμπληρώσουμε και άλλα στοιχεία. Άρα λοιπόν μιλάμε εδώ για ένα τομέα ο οποίο δεν μας δίνει μεγάλες δυνατότητες αλλά θα πρέπει να προβούμε σε βελτιώσεις γιατί πραγματικά θέλουμε μια κοινωνική Ευρώπη και όχι απλά μια Ευρώπη οικονομική διάσταση. Από εκεί και μετά βέβαια θεματοφύλακες τη νομοθεσία τη κοινοτική είναι η Επιτροπή. Και εντάξει, ε, βλέπουμε το τι γίνεται ε, με το, για παράδειγμα με τις ε, καθυστερήσεις των, σε διάφορες πτήσεις οι οποίες προφανώς έχουν και επιπτώσεις σε ό,τι αφορά το προσωπικό που εργάζεται. Έτσι, δηλαδή Ε, τα πράγματα είναι και πολύ πιο σοβαρά. Γιατί άλλο πράγμα είναι να έχω δουλέψει εγώ για παράδειγμα 12 ώρε και εκείνο που μπορεί να μου συμβεί είναι να μου χυθεί ο καφέ και άλλο πράγμα είναι ένα πιλότο να έχει εργαστεί για 12 ώρε. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε ε, τι κάνουμε ακριβώ σε αυτό το επίπεδο. Μετά αποτελεσματικότητα και ασφάλεια. Και η ασφάλεια έχει ε, αντιμετωπιστεί από πλευρά αποτελεσματικότητα και είναι σαφέ εδώ ότι εάν δεν προσφέρω του κατάλληλου μισθού δεν θα έχω και τι κατάλληλε τα κατάλληλα προσόντα, επαγγελματικά προσόντα για το προσωπικό. Δηλαδή, από τη μία προβλήμα σε ντάμπινγκ μισθών, από την άλλη πλευρά προβαίνουμε σε κάποιε ανόητε διαδικασίε ελέγχου, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τα υγρά. Άμα λοιπόν ε, πραγματικά ε, προσλαμβάνονται στα αεροδρόμια άνθρωποι οι οποίοι δεν, είναι, δεν έχουν τα κατάλληλα προσόντα ακριβώ επειδή είναι αναγκαίο να γίνει κάτι τέτοιο, ε, εσεί τι σκοπεύετε να κάνετε. Από εκεί και μετά και η ασφάλιση ασθενεία και γενική υγεία είναι ένα ζήτημα που μα απασχολεί. Για παράδειγμα στην γερμανική τηλεόραση αναφέρθηκε επανειλημμένα πω το, ο αέρας, ο ατμοσφαιρικός αέρας δηλαδή μέσα στην κάμπινα ε, μπορεί να έχει σχέση με καρτινογέννες δηλαδή δεν είχαμε εδώ να κάνουμε με κάποιες ε, κοινοτικές ε, αρχές ή εθνικές αρχές αλλά, οι οποίες προέβησαν δηλαδή σε ένα τέτοιο ε, έλεγχο αλλά ιδιωτικά κάποιοι πιλότοι απευθύνθηκαν σε ιδιωτικές κλινικές και γιατρούς και πράγματι υπήρξε μέτρηση στον αέρα της καμπίνας υπήρξαν κάποιες μετρήσεις οι οποίες έδειξαν πραγματικά ανησυχητικές τιμές εδώ τέτοιων μουσείων ε, και το πρόβλημα αυτό είναι γνωστό εδώ και ε, πολύ καιρό. Ε, μάλλον θα χρειαστεί να περιμένω μέχρι το 2011 ίσως και μετά για να λάβω μια απάντηση από δική σας πλευρά. Σας ρωτώ λοιπόν τι, τι συμβαίνει, γιατί δεν κάνετε ε, τίποτα. Ε, γιατί αν μα λέτε ότι εντάξει θα περιμένουμε άλλο ένα χρόνο και θα δούμε τι θα γίνει και θα πρέπει να το ερευνήσουμε παραπάνω, ε, δεν κάνουμε τίποτα. Δηλαδή πείτε μα, ήταν σωστή αυτή η αναφορά ότι υπάρχουν τέτοιε ουσίες, είναι μολυσμένο ο, αέρα τη καμπίνα ή όχι. γιατί αν ισχύει πραγματικά βάζουμε σε κίνδυνο τη ζωή αυτών των ανθρώπων. Μετά, ένα άλλο ζήτημα που αναφερθήκατε είναι αυτό του, του low cost, δηλαδή την, ε, αεροπορικών εταιριών χαμηλού κόστους. Για παράδειγμα, η EasyJet ε, ε, φεύγει, πετάει από το Σιόνεφελτ προς τις Βρυξέλλε. αλλά άκουσα από πολλούς συναδέλφους ότι συχνά υπάρχουν κάποιες ακυρώσεις πτήσεων και δεν είναι πάντοτε σίγουρο ότι αποζημιώνονται αυτές οι πτήσεις ή κάποια επιχειρήματα δηλαδή ότι υπάρχουν από πλευρά αεροπορικής εταιρείας υπάρχουν διάφορε δικαιολογίε για ε, να μην πληρώσουν και μετά, ε, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά την ευθύνη του για να καλυφθεί αυτή η κατάσταση, για παράδειγμα, δηλαδή να προσφερθεί ένα εισιτήριο από άλλη αεροπορική εταιρεία για αυτά τα άτομα για να μεταφερθούν στον προορισμό του, ε, λένε όχι ότι επειδή είναι ακριβότερα εκείνα τα εισιτήρια δεν είναι δυνατό κάτι τέτοιο, αλλά δεν μπορεί να υπάρχει μια τέτοια εκμετάλλευση. Γιατί πραγματικά, εάν μια αεροπορική εταιρεία κινείται και συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, είναι σαφέ ότι δεν θα σέβεται και κοινωνικού χαρακτήρα σε ό,τι το προσωπικό τη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το θέμα με τις εκθέσεις είναι ότι ιδιαίτερα πλήρης ε, και φαίνεται ότι ε, δεν έχουμε τι να πούμε και μπορώ να σας πω ότι είναι πάρα πολύ πολύπλοκα τα πράγματα. Καλωσορίζω την έκθεση και ακόμη και αν ε, και έχουμε δυσκολίες συλλογής δεδομένων κατά αυτή τη δεκαετή περίοδο, νομίζω ότι γενικά αποτελεί μια καλή σύνοψη σε σχέση με το πώς κινεί το κλάδος. Αλλά θα ήθελα να σταθώ σε ορισμένα σημεία που τέθηκαν, όπως οι συγχωνεύσεις των εταιριών και όπως ξέρετε, εγώ είμαι ένα από τα που έχει περάσει πάνω από 20 χρόνια στον τομέα αυτός και εγώ άρχισα να εργάζομαι στο τομέα όταν, ε, όταν είχαμε μόνο εθνικές εταιρείες. Πριν πολύ καιρό δηλαδή και τελικά αντί να πετάνε τώρα μόνο οι πλούσιοι και οι οικονομικά ε, εύποροι, τώρα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό του κόσμου μπορεί να κινείται σε όλο τον κόσμο. Και αυτά είναι καλά νέα. Είχαμε ένα εγγραφό, θα θυμάστε, για ε, την ε, παγκόσμια πρόκληση της ενίας αγοράς πριν 8-9 χρόνια και ε, το συμπέρασμα ήταν αν οι παγκόσμιες συμμαχίες ήταν ένα καλό πράγμα και καταλήξαμε στο στη συνασπισμή είναι καλό πράγμα γιατί οι πάρα πολύ μικροί αερομεταφορείς δημιουργούσαν τέτοιες, τέτοιους συνασπισμούς με μεγάλους αερομεταφορείς και έτσι ε, βελτίωναν ε, την κατάσταση και τροφοδοτούσαν ε, τις ε, θέσεις εργασίας και από ό,τι βλέπουμε ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να διασφαλίσουμε ότι θα παραμένουν ανοιχτά τα περιφερειακά μα αεροδρόμια. Έτσι λοιπόν, όταν μιλάμε για αυτού του συνασπισμού. εγώ θα ήθελα να πω ότι ε, υποστηρίζω ε, αυτού του συνασπισμού μεταξύ των εταιριών, όμως το θέμα έχει να κάνει με την εργασία και με τι συμβάσει. Δεν είμαι σίγουρη και να ρωτήσω την Κομισιόν προ τα που οδεύουν τα πράγματα, γιατί εσείς υπογραμμίζετε μία σειρά νομοθετικών εκθέσεων που πέρασαν από το σύστημα όταν μιλάμε για τους μετακινούμενους οργανιζομένους κτλ. Εγώ ειλικρινά σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορώ να δω διαφορά εδώ στους εργαζομένους ε, στις ενέργειες μεταφορές σε σχέση με τους εργαζομένους σε άλλους τομείς. Αν πάω να εργαστώ στη Γερμανία, στην Αμερική για μια εταιρεία βρετανική ίσως, αλλά μπορεί να έχει μια θηγατρική και ένα υποκατάστημα. Ε, πολύ συχνά θα υπάρξουν τοπικές ε, συμβάσεις. Έτσι λοιπόν ε, δεν βλέπω να υπάρχει εδώ τέτοιο θέμα όπως θέσατε. Πόσο γνωρίζω και η ΕΛΕΜ έχει προσωπικό που δουλεύει για αυτή και το προσωπικό για την Air France δουλεύει για την Air France. Δεν μετακινούν το προσωπικό, ίσως να είναι πιο ευέλικτη για τη συντήρηση λόγου χάρη των σκαφών, αλλά γενικά είναι ξεχωριστέ οι εταιρείε και δεν βλέπω να υπάρχουν επιπλοκές. Αυτό που με ανησυχεί όμως κάπως είναι το εξής. Πώς ε, θα το προχωρήσουμε το θέμα αυτό, θα έχουμε κάποια νομοθεσία και θα λάβουμε αποφάσεις για τις εταιρείε. Εμείς ε, ε, θέλουμε να σταματήσουμε τις κρατικές ενισχύσεις αυτές. Οι εταιρείε είναι επίλυσης εμείς ε, είμαστε υπεύθυνοι και τα κρατημένοι είναι υπεύθυνα για θέματα όπως να καθορίζουν τον ελάχιστο μισθό κτλ. Έτσι λοιπόν ε, εδώ με ανησυχείτε ότι θέλουμε να έχουμε διαφορετική μεταχείριση αυτού του τομέα σε σχέση με τους υπολείπους. Είναι πολύ ενδιαφέρον να έχουμε μία συζήτηση, όντω, αλλά αν μου επιτρέπετε να πω και κάτι ακόμη, Πρόεδρε. Όπω είπατε, αναφερθήκαμε σε θέματα εναρμόνιση ε, για το προσωπικό ε, και αναφέρεται και ένα νόρο κλειδί όπως είναι η ασφάλεια. Έχουμε την ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφαλείας και την υποστηρίζουμε και προσπαθούμε να έχουμε εναρμόνιση, είτε μιλάμε για ιδιωτικές εταιρείες, για ε, την κυκλοφορία των επιβατών. Έχουμε πολλά προβλήματα σε αυτό το τομέα. Ένα κύριο πρόβλημα είναι το προσωπικό ε, του αεροσκάφους. Ε, υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλα θέματα στην μέσα γιατί κάποιοι φαίνεται να πιστεύουν ότι είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να υπάρχουν και ε, γιατροί. Όμως, ε, ξέρετε ότι ε, μάλλον να γίνονται εξετάσεις ιατρικές για το προσωπικό, όμως απαγορεύεται να μην απασχολείται το προσωπικό κάθε χρόνιο για κάποιες ε, μέρες και να μην πετάει. Όμως αυτό ισχύει για τις μικρές εταιρείε. όμως πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί για το πού πηγαίνουμε. Έτσι λοιπόν, θα ήθελα να πω ότι καλωσορίζω το εγγραφό σας και καλωσορίζω και το μελλοντικό έγγραφο που θα εκπονήσετε για του χρόνου, αλλά θα ήθελα να είμαστε σόφρονες εδώ. Γιατί καλό είναι να το βλέπουμε το πράγμα συνολικά, αλλά θα ελπίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα παρουσιάσει οδηγίες ή κανονισμούς που θα παρεμποδίσουν την ευρωπαϊκή, τις ευρωπαϊκές να ανταγωνιστούν διεθνώς, γιατί εδώ δεν έχουμε καιρικά φαινόμενα 11 Σεπτεμβρίου, η Φέστο κτλ. Εδώ πρέπει να σκεφτούμε ότι αυτές οι αεροπαρικέ εταιρείε ε, δίνουν θέσεις εργασίας και κέρδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θέλουμε να έχουμε ασφαλείς αεροπορικές εταιρείε και θέλουμε οι εταιρείε μας να μπορούν να ανταγωνίζονται παγκόσμια και όχι το ένα του χέρι να είναι δεμένο πίσω από την πλάτη. Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ πολύ. Δεν ε, βλέπω να έχει ζητήσει κανεί άλλο λόγο. επιτρέπετε να πω δύο λόγια. Πρώτα απ' όλα, να σε ευχαριστήσω για την παρουσίασή σα σήμερα. Φαίνεται ότι ε, εκφράσατε πολλά που έχουμε αισθανθεί και εμείς όσον αφορά την απελευθέρωση τα τελευταία αυτά χρόνια. Ορισμένοι από εμά βρισκόμασταν στο κοινοβούλιο αυτό όταν είχαμε την πρώτη δέσμη μέτρων στον αεροπορικό τομέα και τη δεύτερη και την τρίτη. Το είδαμε να γεννιέται ε, αυτό το θέμα και όπως είπε η κυρία Φώστερ, ξέρετε, αρχικά ε, ήμασταν κατά των εθνικών αερομεταφορέων, κατά των εθνικών ενισχύσεων που κατά κάποιο τρόπο ε, καθιστούν ε, το, τα επαγγέλματα στον τομέα των εμπορικών μεταφορών ως ε, μια, ως μια σειρά από υπηρεσίες ελίτ. Όταν όμως θέσαμε το ερώτημα το κατά πόσον με μια έννοια αυτό το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή ε, ίσως γέρνει από την άλλη μεριά πλέον και πάλι όμως με έλλειψη ισορροπίας. Κατανοώ ότι η απελευθέρωση παρουσιάζει ωφέλη για, το, για τους ταξιδιώτες Τώρα μπορούν ε, οι επιβάτε να μεταβούν εκεί όπου στο παρελθόν δεν θα μπορούσαν. Βέβαια, ορισμένοι περιβαλλοντολόγοι λένε ότι αυτό αποτελεί καταστροφή του πλανήτη. Αλλά αυτό είναι ένα επιχείρημα το οποίο το έχουμε ακούσει και το ακούμε. Εγώ πιστεύω βεβαίω ότι η απελευθέρωση έχει ωφέλη. Και το γεγονό ότι έχουμε τώρα ιδιωτικέ εταιρείε κτλ. Φαίνεται όμως τελικά ότι τους, τους εργαζόμενους δεν τους ωφέλησε στον ίδιο βαθμό. Δέχομαι ότι αυξήθηκε ο αριθμό των ε, θέσεων εργασίας. Όμως όταν μου λένε ότι η απελευθέρωση η περισσότερε θέσει εργασίας εγώ τίνω να είμαι κάπως επιφυλακτικό. Κοιτάξτε, ε, ε, η κατασκευή του αποχετευτικού συστήματος ε, στην, στο Ηνωμένο Βασίλειο δημιούργησε θέσεις εργασίας. Αλλά δεν νομίζω ότι τότε ήθελαν αυτές τις θέσεις εργασίας. Άρα να δούμε και την ποιότητα των θέσεων εργασίας. Και εδώ νομίζω ότι η ποιότητα σε αυτό το πακέτο απελευθέρωσης δεν αυξήθηκε δεν ακολούθησε ε, την ε, αύξηση του αριθμού των θέσεων εργασίας. Οι, οι ποιοτικέ θέσεις εργασίας μειώθηκαν. Άρα δεν ξέρω κατά πόσο ε, ε, ωφελήθηκε το εργατικό δυναμικό από αυτή την απελευθέρωση. Η απελευθέρωση μας έδωσε τη Ryanair, την EasyJet, ορισμένοι θα πούνε «Α, μάλιστα, αποτυχία». Όχι, όχι, εγώ δεν σας λέω κάτι τέτοιο. Αλλά έφερε ταυτόχρονα χαμηλά πρότυπα εξυπηρέτησης σε σχέση με το παλιό παραδοσιακό μοντέλο των αερομεταφορέων. Θέλετε ένα παράδειγμα? Για κοιτάξτε την Αερλίνγκου σήμερα. Και ε, πώς ήταν πριν την Ryanair τότε και τώρα. Τώρα, ε, κατά μια ορισμένη έννοια, δεν διαφέρει ιδιαίτερα από τη Ryanair. Οι μισθοί έπεσαν, κατά την άποψή μου. Επίσης, αυξήθηκε ο φόρτος εργασίας. Το είπατε κι εσείς και το επίπεδο εξυπηρέτησης είναι χειρότερο. Ταυτόχρονα είχαμε αριθμό ρεκόρ νέων αεροπορικών εταιριών. Αλλά ταυτόχρονα και αριθμό ρεκόρ χρεοκοπημένων αεροπορικών εταιριών. Αριθμό ρεκόρ ε, νέων παραγγελιών από τη μια και από από την άλλη ε, αεροπλάνα τα οποία είναι αχρησιμοποιητά. Και τώρα έχουμε αυτά τα απίστευτα σενάρια. Αερο... Αεροσκαφό νέας γενιάς, Boeing 737, που ε, πλέον είναι άχρηστα. Άρα, τι θέλω να πω. Ναι, η απελευθέρωση έχει ωφέλη και δεν το αμφισβητώ. Αλλά νομίζω ότι ε, είναι δίκοπο μαχαίρι. Και αυτό το οποίο θα ήθελα να δω εγώ σε επόμενο βήμα, εκ μέρου τη Επιτροπή, είναι πολύ περισσότερη εργασία follow-up σε επίπεδο κοινωνικών πτυχών. Και το πώ επηρεάζεται το εργατικό δυναμικό. Όχι μόνο ποσοτικά. Ναι, υπήρξε αύξηση των θέσεων εργασία. Ναι, υπήρξε. Αλλά ε, ποιε είναι οι αποδοχέ σήμερα σε σχέση με τις αποδοχές στο παρελθόν. Οι κοινωνικές συνθήκες που διέπουν αυτές τις εργασίες τώρα είναι του παρελθόντος. Και ταυτόχρονα ποιο είναι το επίπεδο εξυπηρέτησης προς τους σήμερα σε σχέση με το παρελθόν. Περιμένω λοιπόν από εσά να πείτε σε τελευταία ανάλυση Πώ θα σημειώσουμε πρόοδο. Καλή αρχή, αλλά τι θα κάνουμε τώρα στη συνέχεια και πώ θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το αποτέλεσμα για να καταλήξουμε σε μια έκθεση που θα καλύπτει ολόκληρο το πεδίο τη εταιρική αγορά και τη απελευθέρωση τη αγορά, γενικά στον τομέα των ευρωπαϊκών μεταφορών, συμπεριλαμβάνοντα και αυτέ τι παρατηρήσει που έκανα. Έχετε πάλι το λόγο λοιπόν, αναφέρομαι σαν εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σα ευχαριστώ, Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είναι σαφές και ίσως θα μπορούσα ε, να εκμεταλλευτώ τα πρώτα λόγια. Διακόπτεται ο μιλητής. Euh, Πρόεδρε, ίσως να ξεκινήσω. Δεν υπάρχει τεχνικό πρόβλημα, ρωτάει ο Πρόεδρος. English Για δοκιμάστε πάλι. Εντάξει τώρα. Πολύ ωραία. Μάλιστα. Λοιπόν, έλεγα ότι πρόεδρε θα χρησιμοποιήσω ειδικά στα λόγια και τα λόγια του κυρίου Γκρός. Απελευθέρωση. Ναι. Βεβαίως. Βεβαίω και πρέπει να συνεχίσει και δεν πρέπει να τίθεται σε αμφισβήτηση, αλλά δεν αποτελεί αυτό σκοπό. Έχουμε την πεποίθηση και άλλο αυτό αποδεικνύει και η έκθεση αυτή, αλλά και άλλε μελέτε που κάναμε, ότι η απελευθέρωση του τομέα των αεροπορικών μεταφορών που στην ουσία ήταν σαφώ ε, τομέας ε, κλειστός, άρα ελιτίστικος. Όλα αυτά λοιπόν και η απελευθέρωση είχαν τεράστιο ωφέλη για του καταναλωτέ χωρίς να έχει τις αρνητικές συνέπειες προς εργαζομένους που θα μπορούσαμε να είχαμε φανταστεί. Αλλά αυτό κατέστη δυνατό μόνο επειδή η απελευθέρωση συνοδεύτηκε από την ε, κανονιστική σύγκληση προς, για παράδειγμα, περισσότερη ασφάλεια. Προς την κατεύθυνση αυτή. Είναι αλήθεια επίση ότι τα ζητήματα τη απασχόληση, τη εργασία, των συνθηκών εργασία, των τομέα των Ευρωπαϊκών μεταφορών μέχρι στιγμής εξετάστηκαν κυρίως υπό το πρίσμα ε, της ασφάλειας. Αλλά εδώ πρέπει να είμαστε διάλεκτοι όσον αφορά την ε, ασφάλεια. Η ισορροπία που πετύχαμε ανάμεσα στην απελευθέρωση και στην ανάπτυξη τεχνικών κανόνων είναι μια ισορροπία που βεβαίως ε, δεν είναι τέλεια και σίγουρα θα πρέπει να συνεχίσουμε να την βελτιώνουμε αλλά υπάρχει και είναι εδώ. Τώρα, ο κύριος Γκρός μου έθεσε ένα συγκεκριμένο ερώτημα, το οποίο αφορά ε, την, ε, ε, την εξυπηρέτηση σε ενδιάμεσους σταθμούς. Να σας πω το εξή και θα είμαστε δυνατόν να ακριβέστερος γίνεται. Ήδη έχουμε ξεκινήσει εργασία στο συγκεκριμένο τομέα και έχουμε ξεκινήσει μία μελέτη η οποία προετοιμάζει την εξέταση της οδηγίας συνδρομή σε ενδιάμεσο σταθμό, τι οποίε τα αποτελέσματα αναμένονται στο τέλο του 2010 αρχέ 2011 στα πλαίσια, στα πλαίσια αυτής της εργασίας οι κοινωνικέ πτυχές θα εξεταστούν και εξετάζονται, χωρίς αυτοβολία αυτό θα γίνει και ε, επίσης ε, θα διαβουλευτούμε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Ε, με, με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Επίση, έχουμε ξεκινήσει και μια διαβούλευση με του πολίτε, η οποία ε, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα μα από το Δεκέμβριο έως το Φεβρουάριο και τα αποτελέσματα επίσης θα δημοσιευθούν ε, στο άμεσο μέλλον. Έχουμε την πρόθεση, συγκεντρώνοντα αυτά τα αποτελέσματα, να τα παρουσιάσουμε σε ένα εργαστήρι που θα οργανωθεί στο τέλος του 2010, αρχές του 2011, με ένα πακέτο προτάσεων νομοθετικής φύσεως ε, για τους αερολιμένες ε, κατά το δεύτερο εξάμεινο του 2011. Αυτό ως προς το χρονοδιάγραμμα. Επίσης, θα υπάρξει ανακοίνωση όσον αφορά το πρόγραμμα δράσης για την ικανότητα και τη χωρητικότητα των αεροδρομίων και ε, κυρίως τρεις ε, νομοθετικής φύσεως προτάσεις, ε, ανάμεσα στις οποίες σας αναφέρω μία πρόταση που αφορά τη συνδρομή σε ενδιάμεσους σταθμούς βοήθεια σε ενδιάμεσου βαθμού. Άρα λοιπόν ήδη έχουμε ξεκινήσει τι προσπάθειε ω προ την πτυχή αυτή και επιτρέψτε μου ταυτόχρονα να απαντήσω στον κύριο Καντράουι ε, που, ε, που, είχε μια, που είχε μια παρόμοια ερώτηση. Λοιπόν, τώρα κατά πόσον θα πρέπει να χαιρόμαστε την εξηγήνωση του τομέα ή να ανησυχούμε. Κοιτάξτε, ο κύριος Γκρόση είπε ότι από, μία, ε, από το κρατικό μονοπόλιο θα πέσουμε στο ιδιωτικό πόντο μονοπόλιο. Δεν ξέρω. Αλλά σαφώς εδώ πρόκειται για μία εξυγίανση του τομέα. Την είδαμε ε, και μία ε, ε, δημιουργία συμμαχιών. KLM, Iberia, British Airways, KLM Air France, Lufthansa, SN Airlines. Συμμαχίες και συγχωνεύσεις. Τα πράγματα εξελίσσονται συμμαχίες. Όλες οι συμμαχίες, το τονίζω, πέρασαν από τον έλεγχο του ανταγωνισμού και στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Νομίζω λοιπόν ότι σε αυτό το στάδιο τουλάχιστον και όπως λειτουργεί σήμερα δεν θα πρέπει να ανησυχούμε για λόγους ε, πολιτικής ανταγωνισμού. Εξελισσόμαστε και αυτό βεβαίως δεν μπορεί να γίνει από την μια μέρα στην άλλη. Από μια αγορά ε, ε, στεγανοποιημένη, κλειδωμένη, έτσι για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, απομονωμένοι προ μια αγορά που με μια ανακαλύπτει του κανόνε του παιχνιδιού που είναι τελείω καινούργιοι. Είναι φυσιολογικό υπό αυτέ τι συνθήκε να υπάρξουν και περίοδοι ε, προσαρμογή. Όλα αυτά μεταφράζονται σε μια κάποια αστάθεια. Είναι φυσιολογικό. Αυτό, αυτά έχει η, ζωή ε, στον τομέα της οικονομίας. Έτσι, αν μου επιτρέπετε να το πω, παρόλο που βεβαίως πρέπει να υπάρχει ένα σύνολο ελάχιστων κανόνων. Για παράδειγμα, η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχθεί το κοινωνικό ντάμπινγκ. Δεν μπορεί, ακόμα και αν δεν έχει αρμοδιότητα. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να ασχοληθεί με του μισθού, ούτε με τα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Δεν έχει το δικαίωμα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορεί να, θα μπορούσε η Ευρώπη να, ε, να, να ε, δεχθεί μια ε, ε, κατάσταση κοινωνικού ντάπινγκ και σε αυτό το και σε άλλου χαμηλού, ε, ε, φθηνή, ε, φθηνή αερομεταφορής έναντι κλασικών αερομεταφοριών. Εδώ έχουμε δύο τελείως διαφορετικά μοντέλα. Ή ίσως, αλλά αυτό το δούμε, το low cost αφορά ε, τις ε, ε, βραχίες αποφάσεις, ενώ οι flag carriers, οι εθνικοί αερομεταφορείς θα ασχολούνται με τις μακρινές αποστάσεις και θα έχουμε και μια διάμεση κατάσταση. Αυτή η εξέλιξη έχει να κάνει με την επιλογή του επιχειρησιακού μοντέλου των, των φθηνών εταιριών. Θέλουν να, ε, να, να αξιοποιούν στο μέγιστο αυτό βαθμό τα αεροσκάφη, άρα ε, βραχίες αποστάσεις ε, ε, και όσο το δυνατόν πιο σύντομες ε, και πιο σύντομη διάμεση Θα δούμε σε ποιο, σε ποιο βαθμό είναι βιώσιμο αυτό το μοντέλο. Πάντως μέχρι στιγμή έδειξε ότι αυτό το μοντέλο σχετίζεται με μια κάποια αποτελεσματικότητα. Βεβαίω, λαμβάνοντα υπόψη ότι δεν, επιτρέπεται, στις, δεν επιτρέπει στι επιχειρήσει που ακολουθούν το μοντέλο αυτό να ε, ε, υιοθετούν το κοινωνικό ντάμπινγκ. Αυτό το τονίζω. Πάντως να σας πω και ε, το λέω σε όλους τους, σε όλα τα μέλη τη που τοποθετήθηκαν στο θέμα αυτό και έχουν δίκιο ότι η απόσπαση των εργαζομένων αφορά και τους μετακινούμενους αλλά και αυτούς που δεν είναι μετακινούμενοι. στο τομέα των αεροπορικών μεταφορών το βασικό πρόβλημα είναι το πρόβλημα ε, και των αποσπόμενων και των ε, εργαζόμενων που έχουν πάει για θέση. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο κανονισμός ε, Ρώμη 1 δίνει μια πραγματική λύση. Να εξηγήσω. Ελεύθερη επιλογή σύμβασης. Αλλά η σύμβαση δεν μπορεί να εμποδίζει τον εργαζόμενο από το να ωφεληθεί από τις ε, ε επιτακτικές διατάξεις της χώρας στην οποία ε, ασκεί τις δραστηριότητες του. Δηλαδή, δραστηριότητες, ε, διατάξεις ε, που έχουν να κάνουν με βασικά σημεία του εργατικού δικαίου, με τους μισθούς για παράδειγμα. Με, η διατάξη λοιπόν μιας ε, συμφωνίας που συνάπτεται ελεύθερα και που ε, ε, παραπέμπει σε λιγότερο ευνοϊκέ ε, συνθήκε από τι συνθήκε του κράτου υποδοχή είναι πλέον παράνομε αυτέ τι συμβάσει. Άρα έχουμε μια σημαντική αλλαγή που οδεύει προ την κατεύθυνση περισσότερη προστασία των εργαζομένων. Τώρα, νομίζω ότι απάντησα εν μέρη στις ερωτήσεις του κ. Ελκαντράουε. Κοιτάξτε, πρέπει να το ομολογήσω. Ήδη σα είπα ότι ε, η εν λόγω άσκηση διέπεται από συγκεκριμένου περιορισμού. Δεν έχουμε ιδιαίτερα αξιόπιστα και ακριβή στοιχεία για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε τον όγκο των. Ε, ε, ε τι ποσό των διαδικασιών συντήρηση που αναθέτουν στου εξωτερικού συνεργάτε εταιρείε. Ξέρουμε ότι υπάρχει το φαινόμενο αυτό, είναι σαφέ, αλλά σε ποιο ποσοστό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το μετρήσουμε. Προσπαθήσουμε να το κάνουμε στα πλαίσια της ε, ε, συνέχειας αυτής της άσκησης. Είπα προηγουμένως ε, ότι έχουμε μία προοπτική αναθεώρηση της οδηγίας για την απόσπαση των εργαζομένων και αυτό το είπα γιατί αυτή η ιδέα περιλαμβάνεται στην κοινωνική ατζέντα στην κοινωνική στρατηγική. Έτσι λοιπόν είναι κάτι που είναι σταθερό. Αν μπορώ να σας το πω με αυτόν τον τρόπο. Έτσι λοιπόν, να με ρωτήσατε αν πέρα από το κοινωνικό δίκαιο που θα εφαρμοστεί και στον τομέα των μεταφορών να έχουμε κατά νου και άλλες πρωτοβουλίες που να αφορούν τις, ε, τους αερομεταφορείς. Ε, όχι είναι η απάντηση. Αν και επειδή αυτό το θέμα το προσεγγίζουμε ε, με, την, με τον ίδιο τρόπο που ακολουθήσαμε και στις θαλάσσιες μεταφορές, αν και λοιπόν ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφαλείας ε, να εργαστεί με του Flight Time Limitation από αυτά τα όρια δηλαδή και να ε, εργαστεί και για τις ε, πιστοποίησεις ε, για το προσωπικό και για τις ιατρικές εξετάσεις. Έτσι λοιπόν, το 2009 ξεκίνησαν διαβουλεύσεις, είναι ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο θέμα τεχνικού χαρακτήρα και η ιδέα είναι όταν ε, η υπηρεσία θα έχει ολοκληρώσει το έργο της ε, και θα έχουμε ε, υλοποιήσει μια τεχνική κοινωνική αξιολόγηση να μπορέσουμε το 2012, γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό νωρίτερα, να υποβάλουμε μια πρόταση προς αυτή την κατεύθυνση, η οποία ίσως θα είχε ως αποτέλεσμα το να τροποποιήσει τους εφιστάμενους κανόνες που περιλαμβάνονται σε έναν ε, κανονισμό ε, που εθετήθηκε πριν από κάποια χρόνια. Εργαζόμαστε λοιπόν επί του θέματος αυτού. Είναι ίσως περιορισμένα τα στοιχεία που σας δίνω, αλλά έτσι είναι. Έτσι λοιπόν ε, πάντοτε λαμβάνουμε υπόψη την πτυχή της ασφάλειας, αλλά θέλουμε να έχουμε και ίδιες συνθήκες ανταγωνισμού σε όλη την Ευρώπη και απόλυτη εναρμόνιση. Έτσι λοιπόν, μέσα από το πρίσμα της ασφάλειας προσεγγίσουμε τα κοινωνικά ζητήματα. Όμως τίποτα δεν είναι προκαθορισμένο στο στάδιο αυτό. Κυρία Έλσνερ. Ναι. Ίσως το προσωπικό ασφαλείας ε, στα αεροδρόμια να μην είναι καλά πληρωμένο. Δεν το ξέρω, αλλά να το παραδεχτώ. Εν τω μεταξύ δεν μπορούμε να αναλάβουμε δράση επί του θέματος αυτό, αλλά αναλαμβάνουμε δράση για τον έλεγχο ασφαλείας στα αεροδρόμια. Και σε σύγκριμα ότι οι έλεγχοι αυτοί γίνονται με πολύ σοβαρό και ακριβή τρόπο και σχολαστικό τρόπο και ενίοτε ανακαλύπτουμε για κάποια προβλήματα λαμβάνουμε τα μέτρα που χρειάζεται έναντι των κρατών μελών και γενικά θεωρώ ότι η ασφάλεια των αερολιμένων στην Ευρώπη διασφαλίζεται κατάλληλα. Τώρα για τις πληροφορίες, για τις θέσεις εργασίας, πόσοι άντρες, πόσοι γυναίκες απασχολούνται, πόσες θέσεις εργασίας είναι επισφαλείς ή όχι, όχι, δεν έχουμε τέτοιες πληροφορίες. Πρέπει να εργαστούμε και από αυτό αναφερθήκατε και στις διαφοροποιήσεις ε, ε, των δικαιωμάτων ε, που υπάρχουν μεταξύ των μετακινούμενων, αποσπασμένων εργαζομένων και πάλι. Ένα τμήμα της απάντησης βρίσκει στον κανασμό Ρομπιένα, αλλά δεν είναι το μόνο. Δηλαδή, έχουμε τώρα καταθέσει μια πρόταση για τη δυνατότητα μεταφοράς των δικαιωμάτων συνταξιοδότησης. Βλέπετε λοιπόν ότι ε, βλέπουμε ότι έχουμε εδώ κάτι που να αφορά τις συνθήκες απασχόλησης. Κύριε Κράμερ. Ναι. Ας πράξουμε έτσι ώστε ε, η εθνική νομοθεσία ε, να εφαρμόζεται. Ναι, εδώ συμφωνώ μαζί σας. Η ασφάλεια είναι ουσιαστικό στοιχείο και η κοινωνική συμφωνία που μεταφέρθηκε στο δίκαιο των κρατών μελών το 2000 για τις ώρες εργασίας ελέγχεται. Συγγνώμη, θα μπορούσα να σας ζητήσω να είστε πιο σύντομος. Συγγνώμη, Πρόεδρε, είμαι πάρα πολύ παθιασμένος για το θέμα αυτό, λέει εκπρόσωπος Κομισιόν. Εξετάζουμε τώρα τι εργασίες γίνονται για το θέμα των κοινογόνων χώρων στον τόπο εργασία. Είμαι έτοιμο να αναλάβω πιο άμεση δράση από αυτόν. Τώρα δικαιώματα των επιβατών. Είναι ένα θέμα επί το οποίο εργαζόμαστε. Γνωρίζετε τη δημόσια διαβούλευση που ξεκίνησε στα τέλη του περασμένου έτους θα υπάρξει και μια ανακοίνωση το φθινόπωρο και ίσως αν ε, πρόκειται για την ακύρωση πτήσεων λόγου χάρη θα έχουμε και μια πρόταση αναθεώρησης του κανονισμού 261. Απάντησα, Πρόεδρε, στις ερωτήσεις. Νομίζω απάντησα και στην κυρία Φώστερ. Τώρα, για να κλείσω. Σημείωσα τις επιθυμίες σας. Ήταν πρώτη μου πρόταση αυτό. Εδώ σας είπα ότι κάνουμε μία πρώτη δοκιμή που πρέπει να συνεχιστεί. Ο χρόνος που θα χρειαστούμε θα είναι ανάλογος με τις απαιτήσει ε, που θα υπάρξουν για τη συλλογή των λεπτομερών στατιστικών στοιχείων. Και τελειώνω, Πρόεδρε. Αναφερθήκατε στο σημαντικό αριθμό χρεοκοπιών αερομεταφορέων που είδαμε τα τελευταία έτη. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό, ξεχωριστό θέμα, ίσως θα επανέλθουμε κάποια στιγμή, όμως δεν είναι παράξενο αυτό, καθώς ε, ο τομέας στο παρελθόν ήταν και σήμερα παράγει ένα αγαθό κατανάλωσης, η γεννητικότητα έγινε ένα ειδικαίωμα, ένα κοινωνικό κεκτημένο και δεν είναι ασύνηθες κάποιοι τολμηροί επιχειρηματίες και οι οποίοι εκμεταλλεύτηκαν την καταργήση των εμποδίων στον τομέα αυτή να πήραν υπερβολικά ρίσκα και να έχασαν τελικά. Είναι αρκετά λογικό. Ουσιαστικά θεωρώ ότι εξομαλύνεται η κατάσταση στον τομέα, πρόεδρε, στον κλάδο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ε, και εμεί από την πλευρά τη Επιτροπή μα αναμένουμε με ενδιαφέρον τη συνεργασία μα ε, για τον 261, ε, του κανονισμό 261. Οπότε. Θα είμαστε έτοιμοι για σας όταν θα έρθετε για μελλοντικέ ε, προτάσεις και αναμένουμε τη συνεργασία μας στο εγγύς μέλλον. Να σας ευχαριστούμε πολύ, πολύ για την ε, παρουσίαση αυτή και για τις απαντήσεις που δώσετε στις ερωτήσεις μας. Το επόμενο σημείο στον ημερήσια διαταξή μας είναι ο προπολογισμό του 2011 και προτού δώσω το λόγο στον εισηγητή μας για τον προπολογισμό επιτρέψτε μου να επενθυμίσω στα μέλη της Επιτροπής πως ε, θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την εκπόνηση του σχέδιου γνωμοδότησης με βάση τη συνθήκη της Λισαβόνας μία μόνο ανάγνωση βλέπετε για τον ε, προβληματισμό κατά συνέπεια για τη δική μας ε, γνωμοδότηση. δηλαδή ότι το σχέδιο γνωμοδότηση που θα εκπονήσουμε εμείς θα πρέπει να προσανατολιστεί με βάση αυτό ότι πάμε για μία ανάγνωση μόνο. Ο ο αρμόδιος εισηγητής, οπότε σου δίνω το λόγο, Ντομενίκα, για το σχέδιο προβλησμού του 2011. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπω υπενθυμίσατε, βρισκόμαστε σε ένα κάπως ιδιομόρφο πλαίσιο τη ενία ανάγνωση και από την αρχή, εξάλλου, μας δυσκολεύει κάπως σε επιχειρησιακό επίπεδο. Εγώ καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω του και τους και όλους εισηγητές, με συγχωρείτε, γιατί ε, ε, συνεργαστήκαμε πολύ καλά. Μπορώ να σας πω ότι ήταν πολύ σύντομες οι προθεσμίες ε, και ήταν δύσκολο να εργαστούμε. Έτσι, λοιπόν, μπορέσαμε τελικά να υλοποιήσουμε έργο σε δύσκολες συνθήκες. Αυτός ο προπολογισμό για τις μεταφορές και για τον τουρισμό. Αυτό το σχέδιο της γνωμοδότησης αποτελεί συνέχεια της πρότασης της Κομισιόν. Λογικά περιμένουμε και τη θέση του Συμβουλίου. Θα επανέλθω στο θέμα αυτό σε λίγο, γιατί ήδη έχουμε τα αποτελέσματα της Κορεπέρ, αλλά τη θέση του Συμβουλίου δεν θα την έχουμε παρά σε λίγες μέρες. Και στο βαθμό που πρέπει να ψηφίσουμε την έκθεση αυτή πριν από τις 8 Σεπτεμβρίου, Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι τα μέλη της Επιτροπής αυτής θα πρέπει να εργαστούν σκληρά κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών και να στείλουν τροπολογίε. Έτσι λοιπόν, να, να σας πω ότι αυτό είναι κάπως πολύπλοκο, γιατί εγώ νομίζω ότι ψηφίζουμε στην Επιτροπή στις 2-3 Σεπτεμβρίου για το θέμα. Και βρισκόμαστε και σε ένα πλαίσιο κρίσης. Έχουμε και τη στεγματική αναθεώρηση της συνθήκης της Λισαβόνας που δίνει πραγματικές εξουσίες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά έχουμε μόνο μία ανάγνωση. Ο προπολογισμό από το οποίο θα εργαστούμε, πρόταση τη Κομισιόν δηλαδή, Να σα ε, υπενθυμίσω ότι και πάλι στο παρελθόν είχαμε παρουσιάσει μια γνωμοδότηση στην Κομισιόν ε, να, λάβει καλύτερη υπόψη τον ε, τομέα των μεταφορών. Ο προπολογισμό λοιπόν που προτάθηκε από την Κομισιόν είναι ένα προπολογισμό ο οποίο γενικά είναι ικανοποιητικό. Αλλά το τμήμα ΑΑ ουσιαστικά δεν θα έχει και πολύ περιθώριο ελιγμών, αν έχει και καθόλου, γιατί μιλάμε για 50 εκατομμύρια ευρώ μάλλον. Έτσι λοιπόν η πρόταση γίνεται να αυξήσουμε ναι, κατά 1,7% τις ε, πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και να μειώσουμε τις πιστώσεις πληρωμών κατά 1,7%. Έτσι λοιπόν ε, είχαμε πάρα πολύ, μια πολύ σημαντική πρόταση για αύξηση 10% στα ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Η ανησυχία που έχουμε είναι εξή, να υπενθυμίσουμε ότι είμαστε σε ένα πλαίσιο κρίση και ότι οι μεταφορές και πιστεύω ότι όλοι θα συμφωνήσετε εδώ στην Επιτροπή αποτελούν ένα πάρα πολύ σημαντικό πυλώνα της οικονομικές δραστηριότητας. Είναι και φυσικός πυλώνας γιατί έχουμε ε, τη μεταφορά των υλικών και των ατόμων που είναι στρατηγική σημασία και παράγει το 10% του ΑΕΠ. Έτσι λοιπόν ε, μπορούμε να πούμε ότι αυτό αποτελεί ένα ουσιαστικό στοιχείο ε, και πολύ σημαντική πτυχή και για το περιβάλλον. Γιατί ξέρουμε ότι οι μεταφορές ε, εμπλέκονται ιδιαίτερα στην κλιματική αλλαγή, έχουν πολύ μεγάλες συνέπειες με μη ευνοϊκή τάση. Έτσι λοιπόν στο πλαίσιο αυτό μας ε, φάνηκε ότι δεν θέλαμε να ασκήσουμε κριτική. Η πρόταση που γίνεται στο σχέδιο γνωμοδότησης που σας έχω υποβάλει είναι, σε γενικές γραμμές, να ακολουθήσουμε την πρόταση της Κομισιόν κυρίως ε, στα σημεία που ενισχύει τις υποδομές, ε, τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών, όμως υπογραμμίζοντας ε, ταυτόχρονα ότι δεν έχουν ληφθεί επαρκώς υπόψη οι οργανισμοί. Ο Οργανισμός για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών, που είναι η υπηρεσία της Κομισιόν και υπόλοιποι οργανισμοί είναι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και ένοπλο ε, σκέλος αν θέλετε του Κοινοβουλίου για να εφαρμοστεί η πολιτική που αποφασίζεται από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Έτσι λοιπόν ε, έχουμε δυσκολίες ε, να αποδεκτούμε ότι συστήνουμε κάποιους μηχανισμούς και στη συνέχεια δεν μπορούμε να τους αναπτύξουμε ούτε να τους εφαρμόσουμε τους μηχανισμούς αυτούς γιατί τελικά το ένοπλο σκέλος μας δεν έχει όπλα. Έτσι λοιπόν η πρόταση που έγινε από την Κομισιόν ήταν ανεπαρκής σε ό,τι αφορά τους οργανισμούς, τους agencies. Γίνεται αυτό το σχόλιο αυτό λοιπόν στην έκθεση και η πρόταση είναι να επανέλθουμε στη θέση της Κομισιόν η οποία ήταν ε, μετρίως αυστηρή αν μπορώ να το πω έτσι. Δηλαδή να υποστηρίξουμε και επενδύσεις ε, στα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορέ και να υποστηρίξουμε νέα προπαρασκευαστική δράση για τι μεταφορές σε κοινοτικό πλαίσιο για τις κρατήσεις και το τεχνίξη στο σύνολο των μεταφορών. Αυτό είναι κατά κάποιο τρόπο σαν να προκρίνουμε τη δυνατότητα των χρηστών να ε, μπορούν να έχουν ε, κάποιες πληροφορίες και δυνατότητα κράτησης για διάφορα μέσα μεταφοράς, διατροπικότητα. Σε ό,τι αφορά τώρα τον τουρισμό, δεν έχουμε ειδικό προπολογισμό για τον τουρισμό και οι προσκευαστικές μας δράσεις έγκυται ε, στην Επιτροπή Ήτρε, στο τομέα της βιομηχανίας, περιέργως, έτσι λοιπόν το συζητήσαμε και σε επίπεδο επιτροπής, ζητήσαμε κάποιες προπαρασκευαστικέ δράσεις. Έχουμε δύο προπαρασκευαστικέ δράσεις για το βιώσιμο τουρισμό και για τον κοινωνικό τουρισμό και θέλουμε να έχουμε δύο προπαρασκευαστικέ δράσεις για τον πολιτιστικό τουρισμό και για τον βιομηχανικό τουρισμό. Έχουμε τα σχόλια της Επιτροπής για αυτές τις προπαρασκευαστικές δράσεις. Έχετε λάβει τα σχετικά έγγραφα. Και σε γενικέ γραμμές η Κομισιόν υποστηρίζει τη νέα πρόταση που υποβάλαμε τροποποιώντας την Σύμφωνα με ε, το interface, τη διεπαφή των πληροφοριών για ε, τις διατροπικές μεταφορές, ε, ουσιαστικά προτάθηκε να έχουμε τρεις γλώσσες. Είναι κάπως περιορισμένο το μοντέλο, θα λέγαμε εδώ από ό,τι φαίνεται η πρότασή μα, ε, θα προκαλέσει πολύ σημαντικέ ε, επιπτώσει και στον προπολογισμό αλλά και στο τεχνικό επίπεδο. Έτσι λοιπόν η Κομισιόν έκανε αυτή την πρόταση και αποφάσισε να ακολουθήσει τι υπόλοιπε προτάσει που έγιναν. Και αν μου επιτρέπετε, Πρόεδρε, εγώ θα ήθελα να αναφερθώ και στι προτάσει της Κορεπέρ, γιατί ακόμη και αν δεν έχουμε τη θέση του Συμβουλίου, την πρόταση του Συμβουλίου, έχουμε μια ανεπίσημη θέση του Συμβουλίου μέσω της Κορεπέρ, και μπορώ να πω ότι πολύ δύσκολο να τις ακολουθήσουμε τις προτάσεις αυτές ε, θεωρώ γιατί ε, μέσω της Κορεπέρ ε, προτείνεται ένα μέρο του προβλησμού και θέλω να υπογραμμίσω τριετινά. Έχουμε σημαντική μείωση για τις πιστώσεις στην έρευνα. Αυτό φαίνεται να έρχεται σε αντίφαση ε, με τους στόχους Ευρώπη 2020 και στον τομέα των μεταφορών. Μείωση σημαντική των πιστώσεων για τους οργανισμούς, agencies, ενώ ζητάμε αύξηση και εδώ θέλω να υπογραμμίσω την πρόταση που μου φαίνεται απαράδεκτη να μειώσουμε τόσο πολύ ε, τις πιστώσεις ε, για το σειροδρομικό οργανισμό που έχει διπενικοποιηθεί. Εμείς ζητήσαμε μια αξιολόγηση. Με πολύ καλά επιχειρήματα, έτσι λοιπόν, πολύ δύσκολα δεν μπορώ να αποδεκτώ αυτή την πρόταση, γιατί μιλάμε για μείωση 10%. Επίσης υπάρχει μείωση για τον οργανισμό για τις θαλάσσιες μεταφορές. Πρώτα έχουμε την έρευνα, δεύτερον ε, τους οργανισμούς, agencies και μείωση τρίτον για τις, ε, τα διευρωπαϊκά δικτύα μεταφορών, 10% και πάλι. Εδώ έχουμε κάποια θέματα που πρέπει να υπογραμμίσουμε. Δηλαδή τις υποδομές, την έρευνα και τους οργανισμούς. Ε, εκεί κάνει προσπάθειες στο Συμβούλιο και κάνει τις μεγαλύτερες περικοπές στις πιστώσεις. Έτσι λοιπόν, να συμφωνείτε, θα πρέπει ε, να τα συζητήσουμε αυτά και με τους κοιόδης συζητητές και να κάνουμε κάποιες προτάσεις τροπολογιών που θα είναι να επανέλθουμε στις αρχικές προτάσεις της Κομισιόν και ακόμη και να ζητήσουμε και αύξηση για τα agencies, για αυτούς τους οργανισμούς. Αυτά, Πρόεδρε. Uh, Ευχαριστώ πολύ, Ντόμινικ. Έξι ομιλητέ έχω στο κατάλογο μου. Ελπίζω να μπορέσουμε να προλάβουμε να ολοκληρώσουμε μέχρι τι 5. Καταρχήν ο λόγο του κύριο Λιμπεράτσκι για την ομάδα των σοσιαλιστών. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να εκφράσω την εκτίμησή μου απέναντι στο πρόσωπο του συγκεκριτή του γιατί πραγματικά η συνεργασία μαζί του είναι πολύ ευχάριστη. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον ίδιο τον προπολογισμό, ε, χαιρετίζουμε τα όσα έχουν περιληφθεί εδώ στην ε, εισαγωγή εδώ, δηλαδή τα όσα εμείς έχουμε προβλέψει για την, ε, από την πλευρά σοσιαλιστική ομάδα, για παράδειγμα ε, σε ό,τι αφορά δηλαδή την επένδυση στις μεταφορές για την αύξηση της κοινωνικής κινητικότητας, δηλαδή και άσκηση των δικών μας βασικών δικαιωμάτων. Και και τρόπους για να ξεφύγουμε από την ε, οικονομική κρίση. Επίση, μα άρεσε ο τρόπο που έχει διαρθωθεί ο υπολογισμό και ο τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται από την πλευρά του εισηγητού. Αυτό σε ό,τι αφορά τα θετικά στοιχεία του, της νομοδότησης. Τώρα όμως σε ό,τι αφορά μια ρεαλιστική αντιμετώπιση, μας ανησυχεί λίγο το γεγονός ότι αυτός ο προβολισμός και η σχετική νομοδότηση είναι ο πρώτος που είναι τόσο ορατός. Άρα λοιπόν δεν ξέρουμε κατά πόσο θα μπορέσουμε να επιδείξουμε κάποια πρόοδο διατηρώντα και το status Ο προπολογισμό δηλαδή ε, καταδεικνύει τα όρια χρηματοδότηση που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση και από την άλλη πλευρά χαρακτηρίζεται από ένα μεγάλο, πολύ μεγάλο ποσοστό σταθερών δαπανών, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για νέες δράσεις, για νέες προσεγγίσεις, που ενδεχομένως πράγματι να μην υπάρχουν τέτοια περιθώρια. Αλλά αυτό που δεν μπορούμε να αποδεχτούμε από την ομοδότηση του κυρίου Ρητιά είναι το εξή. Ε, ε, πρόταση Ε, η ε, πρόταση από τον πλευρά του Κορεπέρ, ε, δηλαδή το μόνιμο αντιπροσώπων του Συμβουλίου, να μειωθεί ο προπολογισμό για ευρωπαϊκά δίκτυα Δηλαδή, εάν θέλουμε να βρούμε τρόπου για να εξέλθουμε από την οικονομική κρίση, δεν μπορούμε να δυσκολεύσουμε τον ίδιο μας τον εαυτό, δηλαδή επιβραδύνοντα, δημιουργώντα εμπόδια στην ανάπτυξη των διευρωπαϊκών δικτύων. Ως σοσιαλιστική ομάδα, έχουμε να πούμε πω ε, εμείς αποτύχαμε σε ό,τι αφορά δηλαδή, και τη σχετική ψηφοφορία που έγινε την περασμένη εβδομάδα ε, στο ε, Στρασβούργο. Η τροπολογία, η περίφημη τροπολογία υπαριθμών 6 ασχολούνταν με α, ακριβώς τα σκονδύλια εκείνα τα οποία που κατευθύνονται σε αλλού εκτός δηλαδή των διαθετικών ταμιουργίων σε ό,τι αφορά τα αντιευρωπαϊκά δίκτυα και δυστυχώς δεν καταφέραμε να περάσουμε αυτή την τροπολογία και να διασφαλίσουμε την αξιοποίηση αυτών των κονδυλίων κάπου αλλού, δηλαδή κονδυλίων τα οποία δεν αξιοποιούνται. Συζητήσαμε όμως ε, την δημιουργία μιας αρχής η οποία θα μπορεί να συντονίζει τα κονδύλια από τις εταιρικές σχέσεις ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, αλλά κάτι τέτοιο ε, θα ε, οργανωνόταν ούτω ή άλλω. Δηλαδή, ε, μια σχετική αναφορά δεν χρειάζεται να γίνει στη συγκεκριμένη γνωμοδότηση. Ένα ακόμα σημαντικό ερώτημα που θέτουμε εδώ είναι η το ζήτημα της agency, της αρχής και ο κίνδυνος να μειωθούν τα κονδύλια χρηματοδότησης της αρχής. Μέχρι στιγμή θεωρούσαμε ότι οι σχετικέ υπηρεσίε, οι σχετικέ αρχέ έχουν καλυφθεί από πλευρά χρηματοδότηση και ήμασταν συχνά κατά τη δημιουργία του, εάν δεν είχαν διασφαλιστεί τα κατάλληλα κονδύλια για τη χρηματοδότησή του. Άρα λοιπόν δεν τίθεται καν ζήτημα για μα ε, περικοπή ε, των κονδυλίων των υπηρεσιών γιατί σε διαφορετική περίπτωση πώ θα μπορέσουν να ανταποκριθούν στις ε, αρμοδιότητε του, στι ευθύνε του, Δηλαδή είτε έχουν λόγο ύπαρξη και θα πρέπει να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένε ευθύνε, είτε όχι και να μην υπάρχουν. Επίσης γίνεται εδώ μια αναφορά ότι ο προπολογισμό βρίσκεται στα επίπεδα που είναι απαραίτητα για να διατηρηθεί ο ρυθμό εφαρμογή τη ευρωπαϊκή πολιτική. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, το 2011 θα είναι ένα ασύνδετο έτο ε, γιατί η δική μας ε, δημόσια πολιτική ολοκληρώνεται ως ε, πολιτική μέσα στο 2010, οπότε σε ό,τι αφορά το ρυθμό εφαρμογής των σχετικών κανονισμών, το 2011 θα συναντηθεί από προβλήματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά κάποιε πρόσφατε εξέλιξει, ε, σε ό,τι αφορά τον Γαλιλαίο, είπαμε ότι πέρασε από τι μεταφορέ στη βιομηχανία και παρότι αυτό συνέβη, ε, τελικά αναρωτιόμαστε αν έχει ή είχε πράγματι να κάνει το Γαλιλαίο με τις ε, μεταφορές και τον τουρισμό, αν είχε να κάνει τελικά με το όνομα ενό συγκεκριμένου επιτρόπου ή όχι. Αλλά εν πάση αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Έτσι έχουν ε, τα πράγματα. Η ικανοποίησή μα λοιπόν με τον προπολογισμό είναι αρκετά περιορισμένη, αλλά ευχαριστούμε παρόλα αυτά τον κύριο Ρουκέ για την κριμοθέτησή του. Ευχαριστώ κύριε Γιάνσεν. Σε ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον κύριο Ρικέ για την εργασία του και εγώ πιστεύω ότι ε, κατέβαλε πολύ ε, εδώ μια πολύ σοβαρή προσπάθεια και βρισκόμαστε σε μια περίεργη κατάσταση όπου το Συμβούλιο φαίνεται ότι δεν είναι έτοιμο να ακολουθήσει ε, ε, τον τρόπο χειρισμού. Αναφέρεται η γραπτή διαδικασία. Θα περιμένουμε για να δούμε τι ψήφισε. Δεν έχουμε λοιπόν τα αριθμητικά στοιχεία του Συμβουλίου ακόμα. Και εγώ πιστεύω ότι βασικά θα πρέπει να στηριχθούμε στην υπόδειξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να γνωρίζει τι χρειάζεται, τι είναι απαραίτητο. Πάντως είναι δύσκολη συζήτηση και η διαπραγματεύση με το Συμβούλιο λόγω των οικονομικών δυσκολιών. Άρα δεν βλέπω ιδιαίτερα αισιόδοξα την περίπτωση να έχουμε χρήματα παραπάνω από αυτά πρότεινε η Επιτροπή. Αλλά νομίζω ότι ε, πρέπει να, εδώ θα μπορούσαμε να δούμε τι γίνεται με, τις, ε, με, με τους οργανισμούς. Ε, νέα καθήκοντα στους οργανισμούς και τελικά έχουμε αυτές τις περικοπές. Βλέπε Γκαλιλαίο. Και βεβαίω θα πρέπει να ε, προβλέπεται η επαρκή χρηματοδότηση για να μπορέσουν οι οργανισμοί να ασκήσουν τα καθήκοντά τους. Τώρα, όσον αφορά τα πιλωτικά σχέδια και τι προπροσκευαστικές δράσει, προτείνουμε διάφορες δράσεις και ιδιαίτερα στο τομέα του τουρισμού. Δεν ξέρω, δεδομένη της κατάστασης στην οποία βρισκόμαστε, μήπως ήταν πιο προσεκτικό, πιο σωστό, να μην έχουμε αυτές τις τέσσερις για τον τουρισμό, δηλαδή συνεχιζόμενη προσκευαστική δράση για τον κοινωνικό τουρισμό, για τον εφόρο τουρισμό και μετά έχουμε κάποια πιλωτικά σχέδια για τον βιομηχανικό τουρισμό, τον ευρωπαϊκό τουρισμό, την ε, τις ε, διαδρομές πολιτικής κληρονομιάς. Δεν ξέρω, γιατί κοιτάξτε, εδώ πρέπει να θέσουμε κάποιες προτεραιότητες. Δεν ξέρω. Ε, τελικά, ε, μήπως πάρουμε πολύ λίγα για κάθε μία από αυτές τις δράσεις. Μήπως θα πρέπει να κάνουμε κάποια επιλογή, λοιπόν. Είναι ενδιαφέρον το πολιτικό πρόγραμμα για αυτή τη διασύνδεση για ενημέρωση ε, στον τομέα των ευρωπαϊκών μεταφορών και στον τομέα των κρατήσεων. Ε, κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι, και θα απαντήσει βέβαια Επιτροπή, ότι σίγουρα θα πρέπει ε, να πάρουμε κάποια χρηματοδότηση για αυτό το συγκεκριμένο σχέδιο, έτσι ώστε οι Ευρωπαίοι να ε, κλείνουν ένα ειστήριο τρένο, θέλετε, για που θα περνά από ολόκληρη την Ευρώπη. Εξαιρετική ιδέα. Και την υποστηρίζω ιδιαίτερα αλλά βασικά συμφωνώ με τον κύριο Ρικέ και αυτό που με απασχολεί είναι το κατά πόσον εδώ έχουμε υπερβολικά πολλές ιδέες και μήπως στην πράξη δεν μπορέσουμε να τις ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ε, κοιτάξτε, ο κύριος Ρικέ ανταποκρίθηκε στην εντολή των συντονιστών όσον αφορά τα πιλωτικά ε, σχέδια, κυρίως ε, ε, για αυτή τη μορφή τουρισμού. Εξ στο πρασίνο τώρα η κυρία Ντουιράν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ εκφράζω την ικανοποίησή μου για αυτό το σχέδιο γνωμοδότηση, του κύριου Ρικέ, και αν θέλετε να κάνουμε τι υποδείξει ή ε, ορισμένε προσθήκε. Όπω και εσεί και εγώ συμφωνώ στο ότι η μείωση του προπολογισμού για του οργανισμού δημιουργεί προβλήματα και κυρίω αναφορά ε, για τον οργανισμό για του αεροδρόμου. Ξέρουμε τι ανάγκε του συγκεκριμένου οργανισμού. Ε, είναι πραγματικά παράλογο να μειώνεται ο προπολογισμό ε, ενώ ε, έχει αυξημένε ανάγκε, αναφέρονται 27,7 ε, εκατομμύρια. Τώρα, όσον αφορά τα ευρώ. Τώρα, όσον αφορά το θέμα τη διατύπωση παραγράφου 4. Στην παράγραφο 4 αναφέρεται όλε τι τυχέ που συνδέονται με την ασφάλεια και εδώ θα μπορούσαμε να προσθέσουμε μια ιδιαίτερη έμφαση για ε, το μέδο των σιδηροδρόμων. Γιατί πραγματικά έγιναν ορισμένα ατυχήματα στον τομέα αυτό. Και ε, γι' αυτό ακριβώ πιστεύω ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε τον προπολογισμό προ τον ε, οργανισμό για του σιδηροδρόμου, γιατί είναι το θέμα τη ασφάλεια. Επίση, εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακο. Στην παράγραφο 5, στην πρότασή σα, μιλάτε για τις δυνατότητες ε, που προσφέρονται για την καταπολέμηση ε, της κλιματικής αλλαγής, θα πρότεινα συγκεκριμένα αριθμητικά στοιχεία, 30% μείωση ε, των εκπομπών διοξείδου του άνθρακος για όλο το, το τομέα και μετά ε, θέλω να συνδέσω την οικονομική στήριξη και, την, και τη συνδέση του περιβάλλοντος και να προσαρμόσουμε τη σειρά των αντιστοίχων παραγράφων. Τρίτον, πιστεύω ότι πρέπει να προσθέσουμε κάτι στις δικές υποδείξεις όσον αφορά τα δικαιώματα των επιβατών και τι ε, ενημερωτικέ εκστρατείε. Ε, κοιτάξτε, επανειλημμένα έχουμε συζητήσει τα δικαιώματα των επιβατών. Και εδώ λοιπόν θα πρέπει να υπάρξει μια υπόδειξη. Για το το, για το, ε, ε, όσον αφορά τα πιο συγκεκριμένα σημεία που αναφέρονται σε παραρτήματα, όσον αφορά τον αεφόρο τουρισμό, εδώ θέλω ε, το θέμα του Δούναβη να παραμείνει στη μερίστη άταξη. Νομίζω ότι είναι πραγματικά σημαντικό ζήτημα και επιμένω σε αυτό. Για τα διευρωπαϊκά δίκτυα συμφωνώ μαζί σας ότι είναι αρκετά δύσκολο να κάνουμε λιγότερα. Αντίθετα θα προσέθετα και μία παρατήρηση έτσι ώστε να δοθεί προτεραιότητα στις ε, υφιστάμενες μεταφορές και στις ε, συνομικέ υποδομές. Γιατί διαφορετικά ε, οι μεγάλες επενδύσεις απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων και δεν μένουν χρήματα για μικροπράγματα τα οποία είναι χρήσιμα. Επίσης υποστηρίζω την έρευνα στον τομέα αυτό της διασύνδεσης για τις κρατήσεις. Και άλλωστε εσείς είχατε πει και το υποστηρίξαμε κι εμείς στα, όταν είχαμε την ηφαιστιακή τέφρα αυτού του ηφαιστείου που δεν μπορώ να προφέρω το όνομα, ακριβώς ζητούσαμε περισσότερη ε, δυνατότητα όσον αφορά τις διάφορες κρατήσεις ε, και διασύνδεση ανάμεσα στους διάφορους τρόπους μεταφοράς. Πολύ καλό το εργαλείο αυτό και από τη σκοπιά των επιβατών αλλά και, στην, ε, και στα πλαίσια της λογικής εναλλακτικών λύσεων ότι υπάρχουν προβλήματα για μια ορισμένη μορφή μεταφοράς. Επίσης, το Γαλιλαίο. Μερικέ φορέ έχουμε αμφιβολίε για αυτή τη σύμπραξη ιδιωτικού δημόσιου τομέα και τον τρόπο λειτουργία. Άρα θα ήθελα περισσότερα στοιχεία όσον αφορά τι προθέσει στο συγκεκριμένο θέμα και τέλος, στι υποδείξει. Ξανα, ε, στο σημείο 1 και εδώ θα μπορούσαμε να προσθέσουμε ότι οι μεταφορέ αποτελούν σημαντικό στοιχείο τη οικονομία ε, ε, με ε, επιφέροντα ισότητα και ισοτιμία για όλου. Θέλω όμω να προσθέσω ε, και κάτι. Ε, δεν είναι μόνο οι χρήσιμε μεταφορέ, αλλά και οι άχρηστε ε, που καταστρέφουν το περιβάλλον και δεν ευνοούν την κινητικότητα και την προσβασιμότητα όλων. Ε, ε, ε, θα μπορούσαμε λοιπόν, για παράδειγμα, να προωθήσουμε τις βίντεο διασκέψεις, τις διασκέψεις, έτσι ώστε να περιορίσουμε τις άσκοπες μετακινήσεις. Αυτά ήθελα να πω και σε ευχαριστώ. Καθώς ο δικός μας καθώς ο κ. και ο ε, δεν είναι εδώ, θα πω εγώ δύο λόγια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Ρικέ για την ε, γνωμοδότηση αυτή και θα ε, συμφωνήσω με τα όσα ανέφερε η κυρία Γένσεν σε ό,τι αφορά την δημοσιονομική κατάσταση στα διάφορα κράτη-μέλη. Θα πρέπει δηλαδή να αντιληφθούμε πώ έχει γενική κατάσταση και να ακολουθήσουμε την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η δική μας πολιτική ομάδα θεωρεί πως δεν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να αυξήσουμε τον προβλεπόμενο προπολογισμό της προβλεπόμενης δηλαδή δαπάνες για τις διάφορες ε, υπηρεσίες. Ε, σε ό,τι αφορά τώρα τα πιλωτικά προγράμματα για το ολοκληρωμένο σύστημα κρατήσεων για όλα τα είδη ε, μεταφορών, πράγματι πρόκειται για ένα πολύ επίκαιρο ζήτημα και θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή τις ε, πολύ ακριβείς και ε, εύστοχες παρατηρήσεις που κάνει σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Πασκουάλ. Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον κύριο Ρικέ για την ε, έκθεσή του. Δεν μπορούμε να μιλάμε θεωρητικά για τον προϋπολογισμό. Λέμε στα ισπανικά, υπάρχει μια έκφραση και λέμε ψίχουλα είναι όμως ε, ξέρουμε ότι ε, πρέπει να θέσουμε κάποιες προτεραιότητες γιατί δεν έχουμε επαρκείς πόρους. Όμως θα αναφερθώ σε κάποια θέματα που μας απασχολούν όλους χρηματοδότητα ή ε, χρηματοδότηση των αντιευρωπαϊκών δικτύων. Ξέρουμε ε, λέει ότι υπήρχε ένα όνειρο των 28 δις, μετά περάσαμε στα 8 ε, εκατομμύρια και μετά είχαμε τα 30 ε, project που τέθηκαν στην προτεραιότητα και τώρα βρισκόμαστε στην πραγματικότητα. Είδαμε ότι έχουμε ε, πολύ λίγους ε, κοινοτικούς πόρους και οι εθνικοί πόροι θα είναι ακόμη πιο λίγοι. Και έτσι λοιπόν, ε, αν κάνουμε περισσότερες μειώσεις εκεί, τότε θα γίνει αδύνατη η κατάσταση, γιατί πραγματικά θα παραλύσουν και βλέπουμε ότι ήδη παραλύουν κάποια έργα τα οποία μας ενδιαφέρουν όλους. Τώρα, να σας πω για τα agencies, για τους οργανισμούς ε, τώρα. Έχουμε δυνατότητα ελέγχου. Στο παρελθόν μας είχαν κάνει κριτική ότι δεν έχουμε δυνατότητα ελέγχου. Τώρα όμως λειτουργούν καλά οι οργανισμοί και πρέπει να χορηγήσουμε τους επαρκείς πόρους γιατί διαφορετικά δεν χρησιμεύουν σε τίποτα. Κάτι ένας έχει εδώ τα υιοθετημένα παιδιά του. Ε, τώρα σε σχέση με τον οργανισμό της ε, ασφάλειας στις θαλάσσιες μεταφορές, εγώ μπορώ να σας πω ότι έχει αναλάβει καθήκοντα πάρα πολύ σημαντικό και ο οργανισμός ε, κάνει πολύ καλή δουλειά σήμερα και αν μειώσουμε τον προϋπολογισμό του τότε αυτό θα είναι πολύ οδυνηρό γιατί ε, πραγματικά θα έχουμε πολύ αρνητικό αντίκτυπο στις στο έργο του οργανισμού. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον ε, τουρισμό. Ε, ο τουρισμός πέρασε ως κοινοτική αρμοδιότητα τώρα μετά την εθέτηση της ε, συνθήκης της Λισαμόνας και μπορώ να σας πω ότι τώρα σε μια εποχή κρίσης είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό αν δεν ε, προωθήσουμε και το τουρισμό πάλι θα ε, παραμείνουμε στα όνειρα. Όμως θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κύριε Ρικέ για, την, για το ρεαλισμό σας. Εγώ νομίζω ότι πάρα πολύ σοβαρές είναι οι προτάσεις που υποβάλλετε. Δεν μπορούμε εδώ να έχουμε δημαγωγικό λόγο. Ε, ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ ο λαός και πολύ λίγη η τροφή. Έτσι λοιπόν πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον κύριο Ρικέ για την εκθεσή του και για τις ε, προτάσεις του. Θα ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις και να αναφέρω και το σκεπτικό μου. Μας ε, είπατε ότι το Συμβούλιο ήδη ε, θέλει να παρουσιάσει μία μείωση και ουσιαστικά ταυτοποιεί τον ε, προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους εθνικούς ε, προπολογισμούς όμως καμία σχέση δεν έχουν ήδη υπήρξε σημαντική μείωση στον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό ο οποίος είχε καθοριστεί πριν 7 χρόνια και έχουμε και μία χειροτερία δηλαδή ότι δεν χρησιμοποιηθεί δεν θα χρησιμοποιηθεί σε επόμενες δημοσιονομικές προοπτικές αλλά θα το 2014 κανείς δεν θα έρθει να μας πει ότι είχαμε κρίση το 2010 έτσι λοιπόν, εγώ θα ήθελα να επανέλθω εδώ στην ε, ουσία τη υπόθεση ότι πρέπει να διατηρήσουμε τους στόχου και τον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί έχει προκαθοριστεί αυτός ο προπολογισμό και δεν ε, ε, υποφέρει ουσιαστικά από τα ίδια πηγενέλα όπως οι εθνικοί προπολογισμοί και γενικά κάθε έθνος βλέπουμε ότι ε, ε, τώρα ε, προβάλλει τις εθνικές πτυχές. Την οικονομική κρίση όμως ε, εμείς θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τον τομέα των μεταφορών ε, για να αναζωογονήσουμε την οικονομία. Και τώρα να περάσω στις συγκεκριμένες, στις συγκεκριμένες πτυχές, να ρωτήσω κύριε Ρικέ για το ΣΕΖΑΡ. Ε, είδαμε ότι αυτό το project ε, το χρειαζόμασταν ε, επιγόντως και μας είπαν κάποια στιγμή ότι υπήρξε παράλυση. Έτσι λοιπόν θα ήθελα να αναφερθώ αυτό το 25 συν 10 εκατομμύρια αρκούν ή πρέπει να ζητήσουμε κάτι παραπάνω. Με ανησυχεί πάρα πολύ το ότι υπάρχει μείωση στον τομέα της έρευνας στις μεταφορές. Σε ό,τι αφορά τώρα τους οργανισμούς, ε, θα ήθελα να δώσουμε έμφαση στο θέμα της ΕΜΣΑ γιατί πολλές φορές ε, ε, είχαμε επιπλήξεις από τα κράτη-μέλη γιατί δεν χρησιμοποιούνταν σωστά το προσωπικό. Τώρα για τα δικαιώματα των επιβατών είπε ο κ. Κάλλας ότι θα υπέρξει μια ολόκληρη εκστρατεία για την βελτίωση των δικαιωμάτων των επιβατών 2011 και εγώ νομίζω ότι πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση και επίση να σας πω ότι θέλω να προσφέρω και εγώ ένα μικρό πιλωτικό project για τον προπολογισμό που είναι το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για την ε, οδική ασφάλεια. Διάφορες οργανώσεις θυμάτων της ΠΟΛ και οι ε, εθνικοί εισαγγελεί για την οδική ασφάλεια θα ήθελαν να μπορούν να συμμετάσχουν και να μπορούν να υποστηρίξουν τα μέτρα του Κοινοβουλίου και θα ήθελαν και να μας συναντήσουν γιατί πολύ συχνά ε, ε, επειδή Έχουμε πολύ μεγάλο κατακαιρματισμό στις ε, συνεδριάσεις αυτών των ενώσεων. Καλό θα ήταν να υπάρχει ένα φόρουμ. Έτσι λοιπόν ε, θα θέλαμε να έχουμε ένα ποσό σε πληρωμές έτσι ώστε να μπορέσουμε να θέσουμε σε λειτουργία αυτό το φόρουμ γιατί εγώ νομίζω ότι θα μας βοηθούσε πάρα πολύ στην εξεύρεση λύσεων και βέλτιστων πρακτικών για να ε, θέσουμε τέλος σε αυτή τη μάστιγα από φροντινωτική ασφάλεια. Κύριε Μάιστα. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, σύντομα εγώ θα αναφερθώ σε αυτή την γνωμοδότηση, γιατί ήδη πήρε εκ μέρου τη ομάδα μα το λόγο η κυρία Γιάννησεν. Ε, να πω και εγώ πω ε, πραγματικά είναι πολύ θετικό, όπω είπαν και άλλοι συνάδελφοι, το ότι έχουμε τα απαραίτητα κονδύλα για αυτό το ολοκληρωμένο το Integrated Booking ε, System, ώστε πράγματι να ολοκληρωθεί στην πραγματικότητα η ενιαία αγορά. Και ο συνάδελφο, ο κ. Πρόεδρε, μίλησε ε, για την ε, πραγματική αντιμετώπιση, αν θέλετε, σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό. Για παράδειγμα, σε σχέση με τα διευρωπαϊκά, ε, τι είχαμε αναφερθεί ω προ το τι ακριβώ μπορούμε να κάνουμε για να τα εξελίξουμε περαιτέρω και εάν θα είχε νόημα να έχουμε ένα συγκεκριμένο ενιαίο ταμείο το οποίο θα χρηματοδοτεί όλα εκείνα τα έργα τα οποία επιθυμούμε και ρίχνοντα μια γρήγορη ματιά στον προπολογισμό, είδαμε ότι κάτι τέτοιο είναι αδύνατο. Ε, στη Σαραγώσα είχαμε πει ότι ενδεχομένω θα μπορούσαμε να έχουμε μια εράρχηση των προτεραιοτήτων σε ό,τι αφορά τα προγράμματα που θέλουμε να προωθήσουμε. Αντιλαμβάνομαι βέβαια ότι είναι δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Ε, γιατί βέβαια θα πρέπει κάποιο να κληθεί να λάβει αυτή την απόφαση με αποτέλεσμα εκείνοι των οποίων τα έργα δεν θα ε, εγκριθούν να έχουν παράπονα. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο ε, που θα πρέπει να κάνουμε είναι να δώσουμε προτεραιότητα σε διευρωπαϊκά ε, προγράμματα και να τα χρηματοδοτούμε μόνο στο βαθμό που μπορούμε. Ε, βέβαια, δεν είναι πολύ θετικό κάτι τέτοιο, αλλά θα πρέπει να κινούμαστε με βάση τα κονδύλια που έχουμε στη διάθεσή μα. Και πράγματι, σε ό,τι αφορά τον τουρισμό, όπω σωστά υπόθηκε, έχουμε κάποιε νέε αρμοδιότητε εδώ και γι' αυτό θα πρέπει να εκκινήσουμε ένα νέο πρόγραμμα, για παράδειγμα, όπω αυτό του Industrial Heritage, δηλαδή τη κληρονομιά αυτών τον κλάδο και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε από την πλευρά μας εδώ. Ευχαριστώ. Ο κύριο Γκρός. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ε, συνάδελφο. Δεν θα ήθελα να επαναλάβω τα όσα αναφέρθηκαν, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα TNT. Ε, ε, βεβαιώνω και εγώ τα όσα υπόθηκαν. Σε ό,τι αφορά τα agencies, ίσως θα πρέπει να έχουμε έναν διαχωρισμό μεταξύ της λειτουργίας αφενός και των αρμοδιοτήτων αφετέρου. Εάν δηλαδή πραγματικά έχουμε μια υπηρεσία η οποία λειτουργεί ε, με συγκεκριμένο τρόπο και με σωστό ε, τρόπο, αλλά χρειάζεται περισσότερα ε, κονδύλια, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα ότι ενδεχομένω σε μια τέτοια μελέτη να μην είναι αληθή. Τώρα, με βάση την ε, συνθήκη τη Λισαβόνα μπορούμε να έχουμε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο ε, στον προπολογισμό ε, για τον τουρισμό. Αναρωτιέμαι γιατί όχι. Αντιλαμβάνομαι ότι στον προηγούμενο δεν μπορούσαμε να το κάνουμε γιατί δεν ήταν γνωστό ακόμα, δεν είχε ξεκαθαριστεί αν θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά τώρα γιατί να μην το κάνουμε. Επίση, την τελευταία τρίτη ενημερώθηκα σε σχέση με την τροπολογία 6 του κυρίου Λιμπεράτσκι και τα όσα συζητήθηκαν σε σχέση με αυτή. Ε, πάντως ε, πραγματικά ε, ε, σκέφτομαι ότι ίσως στο μέλλον να χρειαστούμε ένα ταμείο μεταφορών. Και δυστυχώς χωρίς μικρόφωνο ο μιλητής. Um, Προσπάθησε το άλλο μικρόφωνο. Πράγματι, έχουμε προτείνει μαζί με τον κύριο Ρικέ τι συγκεκριμένε γραμμέ του προπολογισμού και έχουμε συμφωνήσει σε σχέση με αυτό, αλλά ίσω θα μπορούσαμε να αναφέρουμε στην δική μα αγνομοδότηση ότι ειδικότερα στου τομεί εκείνου στου οποίου υπάρχει έλλειψη πόρων, ε, θα πρέπει οι επιλογές που θα κάνουμε εκεί να γίνονται με μια συγκεκριμένη συνοχή και να μην αναφέρουμε ενδεχομένω ε, το ε, Ταμείο Μεταφορών, αλλά πρόταση διατύπωση συγκεκριμένα να κάνουμε μία ε, παρατήρηση. Η, δηλαδή η δική μου πρόταση διατύπωση συγκεκριμένα να λέει ότι θα πρέπει να γίνει μια βελτιωμένη αξιοποίηση των κοινωτικών πόρων για την προώθηση της καλύτερης βελτιωμένης κινητικότητας για την καλύτερη αξιοποίηση των σχετικών πόρων. Ευχαριστώ. Πριν δώσουμε το λόγο στην Επιτροπή, να σας πω και εγώ το εξής. Πρώτα απ' όλα πιστεύω ότι ο συζητητής έκανε εξαιρετική δουλειά εδώ και μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα πολύ δύσκολο θέμα. Άρα λοιπόν επιτρέψτε μου να συγχαρώ τον κύριο Ρίκε για την εργασία του. Γιατί η έκθεση του χαρακτηρίζεται από την ισορροπία. Λαμβάνει υπόψη με ρεαλισμό την οικονομική κατάσταση, λαμβάνει υπόψη τις απαιτήσει των πολιτικών ομάδων, και κοιτάξτε, ορισμένοι λένε ότι θα πρέπει να έχουμε το Α, θα πρέπει να έχουμε το Β έργο. Α, και επί τη ευκαιρία σα λέω ότι αυτή είναι η δική μου προτίμηση. Ε, μα αυτό διαρκώ συμβαίνει, έτσι. Αλλά να σα πω ότι ε, άμα δεν ζητήσει κανεί, δεν πρόκειται να, να πετύχει και τίποτα. Και σίγουρα η εμπειρία μου με αυτού του προπολογισμού εδώ και πολλά χρόνια είναι ότι άμα ξεκινά με το 10, το συμβούλιο ξεκινάμε με το 5, από το 5 και κάπου στα μισά του δρόμου βρίσκεται η λύση. Άρα, αν ξεκινήσετε από το 5, σα διαβεβαιώ το Συμβούλιο θα ξεκινήσει από το 2. Ε, έτσι έχουν τα πράγματα. Ε, είναι ε, οι πιο σφιχτοχέριδες που έχω συναντήσει ποτέ. Ε, αλλά έτσι είναι οι Υπουργοί Οικονομικών, πάντα έτσι ήταν. Και νομίζω ότι η έκθεση είναι καλή, είναι ισορροπημένη, χαράσει τις προτεραιότητες που εσείς θέλετε ε, στις πολιτικές τους ομάδες και γενικότερα. Και αν θέλετε αυτές τις προτεραιότητες, αν θέλουμε να συνεχίσουμε προς την κατεύθυνση αυτή, τότε πρέπει ε, να ε, ακολουθήσουμε ανάλογη πολιτική. Και αυτό κάνει και η έκθεση. Είναι για πρώτη φορά με το σύστημα αυτό. Δεν είναι εύκολη διαδικασία και προσωπικά πιστεύω ότι ε, ε, ο χειρισμός ήταν καλός. Ε, τώρα να δώσουμε το λόγο στον κύριο Φελίπε από την Επιτροπή. Θα είναι πολύ σύντομο. Πείτε συμφωνεί, ότι άμα αφού συμφωνείτε με το Κοινοβούλιο θα πείτε ευχαριστώ πολύ, λέμε και εμεί ευχαριστούμε και τελειώνουμε. Να, α, σας παρακαλώ να είστε πολύ σύντομο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα είμαι πολύ σύντομο. Ε, να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Ρικέ για την έκθεσή του. Ε, ε, ε, με την οποία συμφωνεί απόλυτα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως έχει. Ευχαριστούμε. Βλέπετε, ευχαριστούμε. Τέτοια απάντηση θέλουμε πάντα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είδατε τι εύκολο που ήταν. Ευχαριστούμε. Ντομινίκ, θες να πεις, να, να συνοψίσεις εν συντομία και μετά να προχωρήσουμε. Ναι, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, Πρόεδρε. Απλά και μόνο ήθελα να κάνω τρεις παρατηρήσεις και να απαντήσω στην συντομία σε ορισμένε ερωτήσει. Πρώτα απ' όλα, να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά όλου του συναδέλφου με του οποίου ε, συνεργάστηκα ε, και τους κοιόδης. Πρώτα απ' όλα νομίζω ότι ε, ε, όλοι έχουμε πιστεί για τη σημασία των μεταφορών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Διαφορετικά δεν βρισκόμαστε και εδώ σήμερα, σε αυτή την αίθουσα. Άρα υπερασπίζουμε την ιδέα ότι η προσθέμενη αξία του τομέα των μεταφορών θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σε επίπεδο προπολογισμού. Γιατί με αυτόν τον τρόπο μεταφράζεται το πρακτικό ενδιαφέρον του Κοινοβουλίου για το συγκεκριμένο θέμα. Δεύτερον, και εδώ νομίζω ότι επίση συμφωνούμε, ότι τα διευρωπαϊκά δίκτυα αποτελούν ένα, σύστημα, ένα θέμα κεφαλαιόδου σημασία στον τομέα των μεταφορών και των, των υποδομών και των επενδύσεων. Συμφωνούμε νομίζω και εδώ. Και εδώ να ανοίξω μια παρένθεση γιατί αναφέρθηκε επανειλημμένα κάτι. Και θέλω να σας πω ότι εγώ πιστεύω απόλυτα στην ανάγκη ε, της ε, ύπαρξης ενός διευθυντικού ταμείου για τις μεταφορές το οποίο θα μπορούσε να χρηματοδοτείται με διάφορους τρόπους είδαμε πως μόνο και μόνο το απλό ε, θέμα ε, αναφορά σε, ε, στα, ταμεία συνοχής δημιούργησε πρόβλημα όχι μόνο σε παιδοέλκα αλλά γενικά. Άρα λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει ε, να ασχοληθούμε με αυτό πολύπλοκο ε, αλλά πρέπει να το δούμε. Πρέπει να δούμε πώ θα οργανώσουμε καλύτερα τα ταμεία συνοχή, έτσι ώστε να υπάρξει ευρωπαϊκή προστέμενη αξία, γιατί περί αυτού πρόκειται, και ίσω να βρούμε και, και ε, ε, νέου πόρου χρηματοδότηση. Είναι πολύ σημαντικό το ζήτημα αυτό ε, και σίγουρα θα υπάρξουν δυσκολίε ε, με την Επιτροπή Προπολογισμού, με την Επιτροπή Ανάπτυξη ενδεχομένω κτλ. Και τρίτον, να σας πω ότι ε, όσον αφορά τους οργανισμούς, οι οργανισμοί πάντα σε γενικές και σε γενικές γραμμές αποτέλεσαν το αντικείμενο υπόνοιας, αν θέλετε. Δηλαδή ότι αποτελούν ένα τρόπο ελέγχου του προπολογισμού και ε, ε, αξιοποίηση του προπολογισμού. Να σα πω ότι όλη η εργασία που έγινε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που συνίσταται στο να υπάρξουν νέε προτάσει, νέα μέτρα, νέοι τρόποι έλεγχη με στόχο και βελτίωση τη λειτουργία τη Ένωση, αλλά και ε, περισσότερη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, όλα αυτά μεταφράζονται σε νέα καθήκοντα για του οργανισμού. Άρα λοιπόν, εάν εμεί δεν ψηφίσουμε και δεν δώσουμε τα μέσα, αν εμεί ψηφίζουμε και δεν φροντίζουμε αυτά που ψηφίζουμε να μπορούν να εφαρμοστούν μέσα των κατάλληλων μέσων, κυρίω σε επίπεδο ε, οργανισμών, τότε δεν έχουν νόημα όλα αυτά. Επανέρχομαι ε, στον οργανισμό του συνοδρόμου. Αν ζητάμε περισσότερη ασφάλεια, περισσότερη διαλειτουργικότητα, περισσότερο άνοιγμα των αγορών, περισσότερε υποδομέ και ταυτόχρονα δεν επιτρέπουμε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για του Συνοδρόμου να εργαστεί προ την κατεύθυνση τη ασφάλεια, τη διαλειτουργικότητα και των συστημάτων ελέγχου, τότε όλα αυτά που ψηφίζουμε και αποφασίζουμε δεν έχουν νόημα. Ναι, να ελέγξουμε του οργανισμού, αλλά να δώσουμε και τα μέσα για να εργαστούν. Αλλά νομίζω ότι σε γενικέ γραμμέ συμφωνούμε όλοι στο συγκεκριμένο ζήτημα. Ε, Δύο-τρει σύντομε απαντήσει που ετέθησαν. Σεζάρ. Προ στιγμή μιλάμε για πιστώσει έρευνα και ε, ε, λυπάμαι που υπάρχει αυτή η, αντιμετώπιση όσον αφορά τις πιστώσεις ε, έρευνας, κυρίως γιατί έχουμε να κάνουμε και με την ασφάλιση των των αεροπορικών μεταφορών και με τα δικαιώματα των ε, επιβατών έμεσα, γιατί αυτά έχουν να κάνουν και με την ασφάλεια. Και επίσης, ε, όσον αφορά τα δικαιώματα των επιβατών και μείωση του προπολογισμού προ την κατεύθυνση αυτή, νομίζω πρέπει να το συζητήσουμε και με το Συμβούλιο και με την Επιτροπή για να δούμε ποιε είναι οι προθέσει του. Σημείωσα το Ευρωπαϊκό Σχέδιο του Φόρουμ για την Ασφάλεια, αλλά δεν είδα να το προτείνεται από το έλεξη επίπεδο συντονισμού. Α, ναι, υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα, πρέπει να το ξανασυζητήσουμε. Μα νομίζω ότι πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να οργανωθούμε. Πάντως νομίζω ότι η ασφάλεια είναι σημαντικό θέμα. Το θέμα της χρονιάς, τουλάχιστον σε επίπεδο ευρωπαϊκής προεδρίας. Και τώρα τελειώνω, αναφέρομαι στην τελευταία ερώτηση γιατί δεν υπάρχει ε, ε, ε, στο δικό μας προπολογισμό ξεχωριστό κεφάλαιο για τον ε, τουρισμό, γιατί αφορά άλλη επιτροπή, άλλον επίτροπο. Κοιτάξτε, εγώ σας το λέω με κάθε ειλικρίνεια. Και με την ιδιότητά μου του νέου μέλους. Εδώ πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και αν πρέπει να υπερασπίσουμε τα πράγματα. Γιατί έχω την εντύπωση ότι ορισμένε φορέ οι μεταφορέ εστιάζουν σε καινούρια ε, θέματα και καλά κάνουν, αλλά δεν ασχολούμαστε με θέματα τα οποία μα αφορούν ε, και μα θίγουν άμεσα. Π.χ. τουρισμό και, και γενικότερα θέματα γενικού ενδιαφέροντο. Και εδώ μερικέ φορέ ε, δεν δίνουμε τη σημασία που θα έπρεπε. Ο τουρισμό, ε, εδώ υπάρχει θεσμικό θέμα. Ή είναι, θέμα, είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής μας, άρα ε, πρέπει να δούμε το θέμα των κονδυλίων και των πιστώσεων σε επίπεδο επιτροπή και αφορά γενικότερα τη λειτουργία του Κοινοβουλίου. Βεβαίω εδώ μιλώ για θέματα που ξεπερνούν τι δικέ μου αρμοδιότητε. Τελειώνω, ε, Πρόεδρε. Βλέπω ότι είμαστε ιδιαίτερα ενωμένοι όσον αφορά την πράσινη των μεταφορών και την καλύτερη αντιμετώπιση, δημοσιονομική αντιμετώπιση του θέματο αυτού, λαμβάνοντα υπόψη τι αντιπροσωπεύει και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σα ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Ρικέ. Προθεσμία για 23 Ιουλίου. Ψήφο στην Επιτροπή Μεταφορών 2 Σεπτεμβρίου. Προ ενημέρωσή σα, ψηφοφορία στην Επιτροπή Προπολογισμού 28-30 Σεπτεμβρίου και στην ψήφιση του προπολογισμού ε, στην Ολομέλεια Οκτώβριο 2010. Θυμάστε όλοι περιμένουμε υπομονησία αυτές τις 4-5 ώρες. Λοιπόν, αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα. Σας ευχαριστώ. Θεωρούμε ότι έληξε η συνεδρίαση. Πριν όμως ε, διακόψω τη συνεδρία, να σας πω ότι αύριο το πρωί θα είμαι εδώ, δεν θα είμαι εδώ, ε, γιατί ε, η κόρη μου αποφυτά δεν θα είμαι εδώ, αποφυτά αύριο την Τρίτη, δεν θα είμαι εδώ, γι' αυτό θα έχετε αύριο τον Αντιπρόεδρο. Καλές διακοπές, ελπίζω να σας δούμε όλους ξεκούραστους και φρέσκους φρέσκους το Σεπτέμβρη. Σας ευχαριστώ όλους. Ναι, στον αθλητισμό ε, σπουδάζει θέματα αθλητισμού. Δεν ξέρω, μπορεί να σα δημιουργεί